Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Κάποια τυπικά διαδικαστικά πρώτα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε την ημέρησα διάταξη. Γίνεται μάλιστα αναμετάδοση της συνεδρίασής μας και διαδικτυακά και δεν έχουμε ε, διερμηνία στα τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και ιρλανδικά. Λυπούμε γι' αυτό. Θα ήθελα παρακαλώ να εγκρίνουμε για τα πρακτικά των συνεδριάσεων 27η 27-28 Φεβρουαρίου και τη κοινή συνεδρίαση της 28 Φεβρουαρίου με την Επιτροπή Γυναικών. Είχαμε συζητήσει στην κοινή αυτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας την έκθεση πρωτοβουλίας για το ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Σίγκβριτ Μούρεσαν, τον οποίο και καλωσορίζουμε εγκαρδιότατα. Είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 και μάλιστα το συγχαίρομαι που ανέλαβε τόσο σημαντική έκθεση και το καλωσορίζουμε θερμά στη σημερινή συζήτηση. Χαιρόμαστε που ήρθατε εδώ κυρία Μούρεσαν για να ακούσετε και τις απόψεις των μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Όπως ξέρετε, ο Τιμπορ Σάνι είναι ο δικός μας συγητής, παρίσταται και ο κύριος Σάνι, Το καλωσορίζουμε θερμά και εκείνον, και θα ήθελα να κάνουμε την εισαγωγή στο θέμα αυτό με την ενημέρωση από το δικό μας συγκεκριτή, τον κύριο Σάνι, που είναι ο πλέον αρμόδιος ε, για να μας κατατοπίσει και μετά θα δώσω το λόγο στον ε, Γενικό Εισηγητή για τον Προπολογισμό, τον κύριο Μούρεσαν. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε την ενημέρωση από τον κύριο Σάνι Τιμπορ, τον Εισηγητή της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω λεπτομεριακά. Πρώτα απ' όλα όμως να καλωσορίσω θερμά τους συναδέλφους και κυρίως τον κύριο Σίκφριτ Μούρεσαν και να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις απόψεις Επιτροπής Γεωργίας εξού και η συμμετοχή σας εδώ σήμερα. Σίγουρα ο προπολογισμό είναι πολύ σημαντικό και ο προπολογισμό τη Γεωργία επίση πολύ σημαντικό, αλλά ιδιαίτερα είναι επίκαιρο αυτό τον καιρό και για πολλούς και διάφορους λόγους ε, θα είναι προτεραιότητα ο γεωρικός προϋπολογισμός ε, στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας εξηγήσω εντός ολίγου γιατί. Ζίκφριντ, σε σένα κυρίως απευθύνομαι ε, και μπορώ να σου πω ότι εκπροσωπώ ήδη και αρκετούς συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας γιατί Είχαμε ήδη λάβει το πρώτο κύμα των ε, σχολείων και παρατηρήσεων από τους συναδέλφους. Κάτι που δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει το θέμα του προϋπολογισμού και κυρίως ε, του γεωργικού προϋπολογισμού στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος ε, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης είναι σημαντικός για την υλοποίηση πολλών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρω και στη γνωμοδότησή μου, ε, έχουμε ένα κατάλογο που μπορεί κάλλιστα να διευρυνθεί, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα θέματα που θα πρέπει να φροντίσουμε, για τα οποία θα πρέπει να μερινήσουμε. Έχουμε λάβει μέχρι στιγμής 67 τροπολογίες, όλες ε, με πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το σχέδιο γνωμοδότησης Επιτροπής μας περιλαμβάνει και κάποια νέα στοιχεία που θα πρέπει να εφαρμοστούν, όπως η μνήα στη ρήτρα του ενεργού γεωργού της ομάδας οργανώσεις παραγωγών, την καταπολέμηση των αθέμετων εμπορικών πρακτικών και την λεγόμενη έξυπνη προσέγγιση για την Ήπεθρο. Στη γνωμοδότησή μας καλωσορίζουμε τα νέα παρατηρητήρια της αγοράς και επισημαίνουμε τη σημασία που έχουν οι δράσεις στον κτηνιατρικό τομέα και στα φυτοϊγειονομικά μέτρα. Γιατί τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε ότι λάβαμε πολλούς ε, ε, αρνητικούς ιονούς στα θέματα κτηνιατρικής προστασίας και το φυτιογειονομικής προστασίας ε, στην Επίρό μας. Επίσης, η κατάσταση της, της αγοράς είναι ένα θέμα που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής. Στην Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, ασχολούμαστε με το θέμα της μεγάλης διακύμανσης των τιμών, της μεγάλης αυστάθειας των τιμών. Και μπορώ να σε διαβεβαιώσω, Ζίγκφριτ, ότι το θέμα αυτό της μεγάλης αστάθειας των τιμών είναι πραγματικά το δηλητήριο της ε, ζωής των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιδεινώνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των γεωργών. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να διατρανώσουμε την ε, επιτακτική ανάγκη της διαφύλαξης ε, του γεωργικού προϋπολογισμού χωρίς καμία περικοπή και την ανάγκη των περιθωρίων στο 2, καθώς και, την κρίση, ε, καθώς και του αποθεματικού της κρίσης. Όλα αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε στη γεωργία. Γι' αυτό και είμαστε κατά οποιασδήποτε ανακατανομής κονδυλίων σε άλλους τομείς. Παρά την αντίθετη γνώμη μου μερικών. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω το μεγάλο αριθμό των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων που τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η πλειοψηφία τους πραγματικά αξίζει και χρήζει περαιτέρω στήριξης γιατί όλα αυτά τα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις ε, αφορούν στοχευμένα σχέδια, όπως το σχέδιο για την έξυπνη ανάπτυξη της υπαίθρου, που ε, αποτελεί προτεραιότητα και χαιρόμαστε που το ε, ενέκρινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι έτσι θα μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην μελλοντική μας κοινή γεωρική πολιτική και πολιτική τροφίμων. Θα ήθελα λοιπόν να περιλάβεις ε, τις ιδέες μας από το πακέτο των συμβαστικών τροπολογιών που θα εξετάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Επίσης, θα έχω θα, θα ήθελα να υποβάλω και μια άλλη ερώτηση. Ίσως είναι λίγο πρόωρη βέβαια. Και δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σου ή να πεις τη γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τις ε, περιστάσεις που δημιουργεί το Brexit. Γιατί έχουν εκδηλωθεί φόβοι ότι αν όχι το 2018, πάντως στο μέλλον, το Brexit θα επηρεάσει πολλές, ε, πολλά θέματα της γεωργίας. Φυσικά δεν μπορούσα να είμαι εξαντλητικός, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόλαβα, ακροθυγώς ανέφερα κάποια σημεία. Ε, προσπάθησα να σταθώ στις βασικότερες βασικές προτεραιότητες Επιτροπής Γεωργίας. Μπορεί να μην τα είπατε όλα, αλλά όντως επικεντρωθήκατε στα ουσιώδη για την Επιτροπή Γεωργίας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Σίγκριτ Μούρεσαν, για να μας παρουσιάσει τη δική του θέση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ που με υποδέχεστε σήμερα. Ήταν σημαντικό αυτό αυτή η ευκαιρία συνάντηση το εβδομάδα του Μαΐου, γιατί το Μάρτιο στο Ινολομέλιο υιοθετήσαμε τι κατευθυντήριε γραμμέ με την έκθεση η οποία περιλαμβάνει και τι θέσει του Κοινοβουλίου για τι πολιτικέ προτεραιότητε για τον προπολογισμό του 2018. Στο τέλο Μαΐου η Επιτροπή μα θα ε, καταθέσει το σχέδιο προπολογισμού για την Ένωση για το 2018 και σημαντικό για μένα ήταν να σα ε, υποβάλλω καταρχά τι δικέ μου θέσει ε, για τι γενικέ προτεραιότητε του υπολογισμού του 2018 και κατά δεύτερον να σας ε, ενημερώσω ότι είμαι στη διάθεσή σας ε, και είμαι να υποστηρίξω τους ε, γεωργούς εν ώψη των εξελίξεων που επί παραδείγματι ανέφερε ο Τίμπορ με τις εξελίξεις για τον Brexit και την απτητικότητα της αγοράς και κατά τρίτον επίσης και αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ θέλω να ακούσω τις δικές σας θέσεις για τις συνθήκες που επικρατούν και την ανάγκη χρηματοδότησης των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προϋπολογισμού του 2018. Κατευθυντήρες γραμμές καταρχάς υιοθετήθηκαν ε, στη Σύνοδο του Μαρτίου στο Στρασβούργο με ευρύτατη πλειοψηφία την οποία οφείλω και πρέπει να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας. Είναι πολύ, ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η πλειοψηφία ακριβώς γιατί έχουμε ενωμένη και ισχυρή φωνή στις διαπραγματεύσεις εναντί του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο Επίτροπος Έτιγκερ στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Μαρτίου αλλά και κατά τις συζητήσεις που είχαμε μαζί του στην Επιτροπή των Προπολογισμών επέδειξε πλήρη κατανόηση για τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες. Έπεισε ότι τις αντιλαμβάνεται και ότι είναι επιτεθειμένος να καταθέσει έναν προπολογισμό, ένα σχέδιο προπολογισμού που θα σέβεται τι πολιτικέ προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Δύο είναι οι κυρίες προτεραιότητες που έχω ορίσει. Πρώτον, ανάπτυξη, θέσει εργασίας. Δεύτερο, ασφάλεια των πολιτών. Και γιατί φρονώ ότι πρόκειται για τα δύο ουσιώδη στοιχεία πάνω στα οποία πρέπει να εστιαστεί ο προπολογισμό του 2018, γιατί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών η πιο σημαντική κρίση που αντιμετωπίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η μεταναστευτική κρίση, το προσφυγικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα Διάθετοντα και κονδύλια από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Διαθέσαμε λοιπόν τα ποσά, στο βαθμό που μπορούσαμε να τα βρούμε για να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, το Ταμείο για την Αφρική, η διευκόλυνση για την Τουρκία, το Μαντάτ. Πράγμα απαραίτητο βεβαίω λόγω τη σημαντική ροή προσφύγων, ε, Πράτοντα το όμως ε, λησμονήσαμε ουσιώδεις προτεραιότητες του προϋπολογισμού και η οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί από μόνη της. Γι' αυτό λοιπόν πρώτη μα προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάπτυξη θέση εργασίας, οι επενδύσεις ε, στους τομείς αυτούς που θα ενισχύσουν την οικονομία μας, θα την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική και σε αυτό εννοώ και τις υποδομές, στην καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρηματίες, τους νέους επιχειρηματίες, Ορίζον 2020, δηλαδή κόσμε συνδέοντας την Ευρώπη. Για την δε την ασφάλεια, όπως γνωρίζετε, η, η οικονομική μας πόρη για τους τίτλους 3 και 4 είναι πολύ περιορισμένη. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε με περιορισμένους πόρους να εξασφαλίσουμε κάτι το ικανοποιητικό. Και σε αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες οι αποκεντρωμένες της Ένωσης που έχουν ευθύνε σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών αφενός, αφετέρου θα πρέπει να αναπτύξουμε τη συνεργασία με την Επιτροπή και να δούμε τι σχέδια έχει ως προς την υποστήριξη της έρευνας στην αμυντική βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να στηρίξουμε και την εγγύη μα γειτονία, αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική τη διάσταση, γιατί βέβαια πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών μας. Πέραν αυτών των δύο κύριων προτεραιοτήτων, οι κατευθυντηρίες μου γραμμές για τη γεωργία είναι πολύ σαφείς. Είναι δεδομένο ότι η γεωργία είναι μία από τις κύριες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο λόγω των σημαντικών ποσών που χορηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και πολύ σωστά χορηγούνται, ε, αλλά και λόγω της συμβολής της στην ασφάλεια των τροφίμων και στη διαχείριση της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατευθυντηριέ μου γραμμές λοιπόν πολύ σαφέ. Υποστηρίζω πλήρη υποστήριξη για τους γεωργούς που επηρεάζονται δυσμενώς από την ε, γρήπη των πτηνών, από το εμπάργκο εναντί της Ρωσίας ή το εμπάργκο της Ρωσίας καλύτερα και όλα αυτά τα προβλήματα και ιδιαίτερα ανέφερα βέβαια τι προτεραιότητε αυτές στην Ολομέλεια, ζητήσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθιαρογός στους γεωργούς όταν αυτοί πλήττονται από προβλήματα που αναφέρει και ο κύριος ε, Σάνη, η επιτητικότητα των ε, τιμών και άλλα ζητήματα και οποιαδήποτε άλλη κρίση που ενδεχομένως να έχει συνέπειες για την ασφαλή προμήθεια τροφίμων υψηλής ποιότητας στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπω γνωρίζετε, πέρσι στην Επιτροπή των Προπολογιστών ε, υποστηρίξαμε ρητά την δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην αντιμετώπιση της κρίση του γάλακτο. Και πριν ακόμη να καταθέσει την διορθωτική επιστολή, η Επιτροπή κάναμε και εμεί τροπολογίε από πλευράς Επιτροπή των Προπολογισμών ζητώντα 600 εκατομμύρια ευρώ υποστήριξη στους γεωργού ε, του γαλακτοκομικού τομέα Σα διαβεβαιώ, δε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι την ίδια γραμμή θα ακολουθήσω και για τον προπολογισμό του 2018. Όταν δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση κρίσεω σε κάποιο τομέα, θα είμαστε στο πλευρό σα και θα καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί γρήγορα, με τρόπο πιστικό και με τα επαρκή ε, και απαιτούμενα εκείνα ποσά. Και μάλιστα αυτό αυτό αφορά και την επικοινωνία με τη δική σας την Επιτροπή αλλά και την ε, δική μας ε, κύριε Πρόεδρε, την Επιτροπή των Προπολογισμών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η επικοινωνία, η καλή επικοινωνία. Δείγμα αυτής μου της διάθεσης είναι η παρουσία μου εδώ και είναι πολύ σημαντικό για μένα ως γενικό ε, εισηγητή σε αυτή τη φάση και κυρίω εν ώψη των διαβουλεύσεων που θα ξεκινήσουμε το φθινόπωρο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να έχουμε γνώση και των θέσεων τη Επιτροπή σα και των οικονομικών, των δημοσιονομικών αλλαγών που εντοπίζεται σε σχέση με τον γεωργικό τομέα κατά το 2018 και να είμαστε ενήμεροι για πιθανέ κρίσει ή άλλε εξελίξει. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε λοιπόν σε περιστάσεις κρίσεως, να σταθούμε στο πλευρό των γεωργών, χρειαζόμαστε επαρκές περιθώριο στον τίτλο 2. Και θέλω να είμαι πολύ σαφής εδώ, το απευθύνω προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επταετές πλαίσιο του 2014-2020 συμφωνήθηκε, δεν ήταν γνωστές ε, πολλές από τις κρίσεις ε, που έχουμε εντωμεταξύ αντιμετωπίσει. Είτε πρόκειται για την τρομοκρατία, την κρίση, την προσφυγική, τα θέματα της ασφάλειας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα στους τομείς αυτούς, ναι βεβαίως, αλλά οτιδήποτε γίνει στους τομείς αυτούς δεν θα πρέπει να ε, γίνει εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών, της γεωργίας, της πολιτικής συνοχής, της έρευνας, της καινοτομίας, των υποδομών. Έτσι λοιπόν, έναντι τη Επιτροπή θα υποστήριξω τη θέση ότι χρειάζεται στο σχέδιο του προπολογισμού επαρκέ περιθώριο για τον τίτλο 2, ώστε να έχει περιθώριο να ανταποκρίνεται σε απρόσμενε περιστάσει όπω αυτέ που αναφέραμε νωρίτερα. Και οι δύο πυλώνε βέβαια τη κοινή γεωργική πολιτική έχουν σημασία και οι άμεσε πληρωμέ, δηλαδή που υποστηρίζουν τον γεωργό αλλά ταυτόχρονα και η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε επαρκείς πιστώσεις, αναλήψη υποχρεώσεων δηλαδή, αλλά και επαρκή ποσά για την ε, πληρωμή των ε, λογαριασμών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της υπαίθρου, γιατί η ταχύτητα με την οποία έρχονται προς πληρωμή ε, άλλοι λογαριασμοί από άλλους τομείς Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ξεκίνησε πολύ γρήγορα, αλλά προχωρά η αποπληρωμή πολύ αργά πλέον. Και όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός για το Γεωργικό Ταμείο, για την ε, Γεωργική Ανάπτυξη, ορίζει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις ίδιες διαχειριστικές αρχές από το πολίτες στο νομικό πλαίσιο 2007-2013 και έτσι δεν έχουμε καθυστερήσεις στις πληρωμές όπως ε, αυτές που σημειώνονται στην πολιτική της συνοχής, όπου μόνο σε μικρά ποσά μπορούν να γίνονται οι πληρωμές. Θα εξασφαλίσω λοιπόν επαρκή ρυθμό πληρωμών, υπάρχουν ήδη επαρκή ποσά. Δεν ε, υπάρχει μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσε να αποστείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό του να μην μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς τη είτε προς τους γεωργούς ή άλλους δικαιούχου. Εν τέλει για τα πιλωτικά προγράμματα. Κύριε Πρόεδρε, όπως και πέρσι, θα ετοιμάσουμε μία δέσμη πιλωτικών προγραμμάτων που θα υιοθετήσει και θα προτείνει προς χρηματοδότηση μέσα από τη συνδιαλλαγή του Κοινοβούλιο. Κάθε, πολιτική, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή, κάθε πολιτική ομάδα, αλλά και με μεμονωμένος βουλευτής, έχει το δικαίωμα να καταθέσει πρόταση για πιλωτικά προγράμματα. Προθεσμία για την κατάθεση των προγραμμάτων αυτών ε, στην Επιτροπή των Προπολογισμών, ξέρω ότι την ενήμερη συναδελφέ, αλλά το υπενθυμίζω, είναι ε, έως αύριο, η προθεσμία εκπνέει αύριο στι 12 το μεσημέρι. Όποιο λοιπόν έχει ε, την διάθεση να στείλει ένα τέτοιο σχέδιο πιλωτικό, ας το στείλει στην Επιτροπή μας μέχρι αύριο το μεσημέρι για να τα ε, ενώσουμε σε μία δέσμη και να τα αποστείλουμε στην Επιτροπή για προκαταπληκτική αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι θα είναι πολλά τα αιτήματα. Για έγκριση μπορούμε πάντως να υποβάλουμε μόνο ε, εκείνα τα σχέδια τα οποία έχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προεγκριθεί με βαθμό α ε, ή β. Εκείνα που θα έχουν ε, βαθμό σ, γ ή χαμηλότερο δεν θα μπορέσουν να προωθηθούν. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τους συναδέλφους μέχρι αύριο τις 12 να στείλουν τα, τις προτάσεις τους. Ξέρω ότι είστε ενήμεροι, απλώς σας υπενθυμίζω. Για να αποστείλουμε, όπως είπα, τις προτάσεις για προαξιολόγηση στην Επιτροπή χωρίς την οποία δεν μπορούν να εξεταστούν οι σχετικές προτάσεις. Αυτά, Πρόεδρε, από πλευρά μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Περιμένω να ακούσω τις δικές σας θέσεις. Ναι, ο μπορώ είχε μια ακόμη ερώτηση για το Brexit και δεν πρέπει να τη λησμονήσω. Πολύ σύντομα θα απαντήσω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε ο αντίκτυπος του Brexit στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί το Brexit το 2018 δηλαδή θα είναι η Βρετανία ακόμη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλήρη δικαιώματα και πλήρη υποχρεώσεις Άρα δεν θα υπάρχει αντίκτυπος, θα είναι μηδενικός ο αντίκτυπος του Brexit για το 2018, αλλά και άλλωστε το υπενήχθηκε ήδη ότι βλέπουμε ήδη μια δυστημία στην, ε, στο σύνολο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό ώψη του Brexit. Το βλέπουμε αυτό. Και όπως είπαμε θα είναι ακόμη μέλος του 2018, άρα και θα καταθέτει τη συνεισφορά της ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και θα ωφελείται από αυτόν, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε περαιτέρω κινδύνους για το μέλλον. Και θέλω να επισημάνω το εξής ότι πρώτον στην Επιτροπή των Προπολογισμών κοιτούμε όλο και περισσότερο την πρόταση για ιδίου πόρου. Λέγεται πολύ συχνά ότι πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί του δικού τη πόρου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα, τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από του δικού τη πόρου, από ιδίου πόρου και βεβαίω αν πρόκειται τώρα να εισαχθεί ένα νέο φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και αν αυτό εκπίπτει από την εθνική φορολογία, θα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον πολίτη ότι δεν επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο. Η δική μας λοιπόν η προσέγγιση θα ήταν ε, ένα ποσοστό από φορολογία του εθνικού επίπεδου αυτομάτως να ε, μεταβιβάζεται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ανεξαρτήτως των εθνικών συνεισφορών, αλλά όλα αυτά βέβαια θέλουν πολλή συζήτηση και πάνω απ' όλα με το Συμβούλιο. Αυτό που θέλω να επισημάνω πάντως είναι ότι μεριμνούμε ότι μας απασχολεί πολύ το ζήτημα του, της σταθεροποίησης, μιας ε, πιο σταθερής και αηφορού βάσει για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ώστε κρίσει όπω αυτή του Brexit να μην μα πλήξουν. Βέβαια, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, είδαμε μια ατυχή εξέλιξη. Την εξή. Το 2013 υιοθετήσαμε το πολιτιστικό οικονομικό πλαίσιο για το έτη 2014 έως 2020, όπως είπα και νωρίτερα. Δεν μπορούσαμε τότε να προβλέπουμε όλες ε, τις ε, προσδόκει τις εξελίξεις που έλεγαν μεταξύ χώρα. Όταν έγινε η σχετική διαπραγμάτευση υπήρχε ένα συγκεκριμένο όραμα για το πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο, είχε κάνει τι προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έγινε η αναθεώρηση με τι προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σημαντικό στοιχείο τη ρήτρα ευελιξία. ότι δηλαδή εάν υπάρχει ανάγκη να διατεθούν κατά πιο ευέλικτο τρόπο ή με διαφορετικέ προτεραιότητε τα κονδύλια κατά το δεύτερο ήμιση του, ε, της του πολιτή δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να έχουμε αυτή την ε, ευχαίρεια να το αποφασίσουμε η ε, όροι αυτή λοιπόν ε, προέκυψαν κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής, Κοινοβουλίου. Εμεί κάναμε ότι μερίδιο από τη δουλειά αυτή μα αναλογούσε, δηλαδή οθετήσαμε ταχύτατα τι προτάσει Μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο Συμβούλιο ήταν έτοιμο την προηγούμενη εβδομάδα να πράξει το ίδιο, αλλά παρεμπόδιζε τη σχετική απόφαση για την αναθεώρηση του Ηνωμένο Βασίλειο και παραμένει σε αυτή την εμπλοκή μέχρι τι βρετανικέ εκλογέ. Όπω είπα λοιπόν, δεν επηρεάζει ευθέω τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2018 η συζήτηση για τον Brexit, αλλά η η άρνηση αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου να συμπράξει στη σχετική απόφαση μα δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την αναθεώρηση και την ευελιξία. Και έτσι θα χρειαστούν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία υπό τον ορίζοντα 2020 μέχρι το τέλο του Πουδουπού γιατί βέβαια και το ΕΦΣΥ έχει φέρει τι δικέ του συνέπειε και υπάρχουν και άλλοι τομεί και λόγοι για του οποίου θα χρειαστεί η ευελιξία να διαθέσει χρήματα σε άλλου τομεί. αλλά όλα αυτά παραμένουν τώρα σε εκκρεμότητα μέχρι να, μέχρι να ολοκληρωθούν οι Βρετανικές εκλογέ. Όπω είπα, δεν έχει αντίκτυπο λοιπόν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό το Brexit, αλλά η άρνηση της Βρετανίας να συμφωνήσει στην αναθεώρηση των πλήτων δημοσιονομικών προπολογισμών δεν ε, μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τη διαχείριση του ποδοπού σε συνθήκες που έχουν προκύψει μετά το 2013. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφου. Πολύ το, τα είπατε. Είπατε αυτά από μένα. Μέχρι στιγμής θα έλεγα αυτά από εσά. Τώρα θα έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με υποβολή ερωτήσεων κυρίω. 1,5 λεπτό παρακαλώ θα έχει το καθένα. Πρώτος ο κύριος Μπέλντερ. 1,5 λεπτό επαναλαμβάνω. Eh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουρεσάν και για την εκθεσή σας και την ανταλλαγή απόψεων. Θεωρώ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική της, ε, η πολιτική, η γεωρική πολιτική είναι μια κοινοτική πολιτική η οποία χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προπολογισμό. Βεβαίως τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλες ε, αρμοδιότητες, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση της χρηματοδότησης που υπάρχει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε σχέση με τον κοινοτικό προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Και ο τομέας της γεωργίας αντιμετωπίζει με συνεχώς νέες προκλήσεις και ένας εύρωστος προϋπολογισμός για την γεωργία έχει μεγάλη σημασία για να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τρόφιμα σε επαρκή ποσότητα και ικανοποιητική ποιότητα και βεβαίως να συνεχίσουν να προστατεύουν το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να δείτε τα προβλήματα της γεωργίας και βεβαίως αναμένουμε και την περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Κύριε κύριος Ροπέ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Χαιρετίζω το ότι ήρθαμε τώρα στο σημείο στο οποίο κάθε γεωργός είναι σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπήρχε μία κρίση και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να ανακάμπτουν οι γεωργοί. Το 2014-2015 χάθηκαν πάρα πολλά κονδύλια και μόνο 20% αυτών έλαβε κάποια αντισταθμιστική χρηματοδότηση. Υπήρχε το εμπάργκο με την Ρωσία, υπήρχαν και προβλήματα που έπληξαν την σοδιά μια σειρά κρίσεων και είναι καλό το ότι κάνουμε τώρα κάτι για να αποζημιώσουμε τους ε, γεωργούς για να μπορέσουν να κρατήσουν την επιχείρησή τους αν δεν ε, λάβουν αυτές τις ενισχύσεις θα έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα στο να αναλάβουν οι νέοι αγρότες με τη σειρά τους ε, τις εκμεταλλεύσεις και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως δίνουμε παντού α, ε, ενισχύσεις γιατί οι γεωργοί από μόνοι τους έχουν και πάρα πολύ μικρή δύναμη εμπορική όσον αφορά δηλαδή τις αγορές και το τι μπορούν να κάνουν για να επηρεάσουν τις ε, τιμές θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και δυνατότητα συνεργασία. Η κυρία Ράς Γκαρσία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή του προπολογισμού που ήρθε να μας μιλήσει σήμερα, αλλά εγώ ε, ανησυχώ τα μάλλα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου ε, ο προπολογισμό ε, και πάλι θα υποστεί τις πιέσεις των μεταναστευτικών ροών και κρίσεων. Δεν νομίζω ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχουμε στη Μεσόγειο, ούτε τα άλλα μας προβλήματα θεωρώ ότι δεν θα είναι ε, ευνοϊκό το πλαίσιο και θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και άλλα προβλεπτά προβλήματα γεωργικά, ενώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως το ρωσικό εμπάργκο. Χαίρομαι που είναι, έχει επίγνωση των προβλημάτων ο εισηγητής ο κ. Μούρισαν, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε λόγους ε, να είμαστε ήσυχοι για το μέλλον, γιατί είδαμε και στο παρελθόν ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε γεωργικές κρίσεις και πάντα και κυρίως ο γεωργικός τομέας είναι αυτός που πληρώνει τα σπασμένα όταν ανακύπτει μια επίγουσα ανάγκη στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις ε, πληροφορίες. Βάλατε στην πρώτη θέση την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας είναι δυνατές στην γεωργία και εμείς στον τομέα της γεωργίας είμαστε ένας ε, μεγάλος εργοδότης. Οι επενδύσεις αυτές ε, πάντα γίνονταν στον τομέα της γεωργίας και πρέπει να το έχει αυτό κατά νου η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Μιλήσατε για τις συνέπειες του Brexit, φοβούμαι ότι ε, δυστυχώς θα έχουμε και άλλες ε, τέτοιες παρόμοιες τοποθετήσεις Μεγάλης Βρετανίας για να μπλοκάρει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η παραγωγή τροφίμων, ε, η ασφαλής παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο εγκαιάται η γεωργία μας και θα πρέπει νομίζω να παραμείνουν στον πρώτο πυλώνα στις άμεσες ε, πληρωμές. Και επίσης το μέσο αντιμετώπισης των ε, κρίσεων είναι σημαντικό, τα είπαν και οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα όσα έγιναν στη δικιά μου την ε, περιφέρεια, στην Μπότντζε, όπου πραγματικά οι παραγωγοί φρούτων επλήγησαν από παγετό. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις και θα δείτε οπωσδήποτε και τις δικές μας προτάσεις που ελπίζω να βρουν αντίκτυπο στην Επιτροπή Υπερπολισμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την πληροφορία που μας δώσατε για τους παγετούς και πώς έπληξε τη Γεωργία. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Τιμποσάνη και τον Σίγκφριντ Μορεσάν τους εισηγητές. Χαίρομαι για αυτά τα οποία ακούστηκαν και κύριε Μορεσάν θα μπορούσατε να είστε μέλος ε, της Επιτροπής μας. Ε, δείξατε μεγάλη συμπάθεια για την υπόθεσή μας και πραγματικά πρέπει να προσέξουμε δεν μπορεί μέσω του Brexit και λοιπόν προβλημάτων να χρησιμοποιηθεί ε, και να πληγεί η γεωργία. Είναι ο μόνος ε, κλάδος στην Ευρώπη που είναι κοινοτικοποιημένος. Υπάρχουν ελάχιστα κοινοτικά κονδύλια και αν σκεφτούμε γιατί δίνει η Ευρώπη 40%-38% του προπολογισμού τους για 14 εκατομμύρια γεωργούς. Κοιτάξτε, πρέπει να τα δούμε τα πράγματα σχετικά. Δηλαδή πρόκειται για το 1% των δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη, για 14 εκατομμύρια γεωργούς που φροντίζουν ε, να έχουμε ασφαλή τρόφιμα και δημιουργούν ε, πάνω από 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ε, Ευρώπη, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το τόσο τραγικό. Και νομίζω ότι μπορεί να σταθεί να συζητήσουμε αν η χύψη δαπάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα των γεωργών. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ απόλυτα με μερικές σκέψεις των παραλληλισάντων. Θα πρέπει να διατηρήσουμε έναν ισχυρό και κατάλληλο προϋπολογισμό ε, επαρκή για να αναγνωρίσουν το ρόλο που οι μικρομεσαίοι γεωργοί ε, διαδραματίζουν στην κοινωνία και τα ωφέλη που προσφέρουν. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός άμεσων και άμεσων θέσεων απασχόλησης που προέρχονται από τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, φυσικά συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε σημαντικά κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον προϋπολογισμό μας αναθεωρήσουμε τις πολιτικές μας για να αποφύγουμε, να προλάβουμε τις κρίσεις, γιατί έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την αστάθεια των τιμών, τις μεγάλες διακοιμάσεις, τις ε, ε, κατακόρυφες πτώσεις των τιμών λόγω της απελευθέρωσης. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε, να μας βάλουν σε σκέψεις και να ε, δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τις αγορές και τις παραγωγές γιατί έτσι αποφύγουμε κάποιες κρίσεις. Τώρα, για τις ε, αναπόφακτες κρίσεις, αυτές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και εκεί θα μπορούσαμε με μια αλλαγή του μοντέλου της γεωργίας ε, να μετριάσουμε αυτές τις κλιματικές αλλαγές και να αποφύγουμε ή να μετριάσουμε τις ε, συναφείς με αυτές τις κρίσεις. Πάντως χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη προς τη γεωργία προς το παρόν. Στη Γαλλική, για παράδειγμα, η παγετή της τελευταίας εβδομάδας προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στα γεώμηλα, ε, σε φρούτα όπως το κίβι, τα κτηνίδια, αλλά και στα αμπέλια. Και από τις πέντε γεωρικές ενδείξεις που έχουμε στη Γαλλικία, ε, τέσσερα προϊόντα έχουν πληγεί, προϊόντα που καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις ε, και αυτές σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στους παγετούς προηγούμενες εβδομάδες και άλλες κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε αρκετά κονδύλια για να λάβουμε υπόψη και αυτές τις, αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Τιμπόρ Σάνι που παρουσίασε πολύ εύστοχα τα αιτήματα της Επιτροπής Γεωργίας για τον προϋπολογισμό και να ευχαριστήσω και τον Σίγμοντ Μούρεσαν που φαίνεται ότι αφογκράστηκε τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί πραγματικά η κοινή γεωργική πολιτική είναι η πιο ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και χρειάζεται έναν επαρκή προπολογισμό εφάμιλο της σημασίας της. Σε άλλες ε, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα η στήριξη, η στήριξη της γεωργίας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωργία δεν είναι μια συνήθις δραστηριότητα. Υπόκειται σε πολλές κρίσεις, αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Φυσικά έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές και δεν επλήγησαν τα προφορά δέντρα μόνο στη Γαλλική και στη Γαλλία το ίδιο. Και την τον Ιούλιο θα έχουμε μεγάλες κρίση, μεγάλη κρίση και προβλήματα στην Και επίσης είχαμε θανατώσει και εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, πτηνά ε, για να περιορίσουμε τη μετάδοση της γρήπης των πτηνών. Και πέρυσι βέβαια αφιερώσαμε 500 πλέον εκατομμύρια ευρώ για να μετριάσουμε κάπως την κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα, αλλά οι κρίσεις επαναλαμβάνονται συστηματικά και έχουμε μεγάλη αστάθεια των τιμών, ενώ στερούμαστε το μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε τέτοιε κρίσει. Και οι ε, συμπολίτε μα περιμένουν πολλά από τη γεωργία, αλλά και από τον αγροτικό κόσμο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία που έχει η ύπεθρο λοιπόν και σίγουρα να μην περικόψουμε το γεωργικό προπολογισμό γιατί έχουν μεγάλε προσδοκίε οι πολίτε από αυτόν. Και μην ξεχνάτε ότι οι γεωργοί αρχίζουν και ξανίστανται και ίσω εξωθηθούν σε ε, στο να ψηφίσουν ακραία κόμματα. Να μην το ξεχνούμε και αυτό. Κύριε Αγγιλέρα, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών, τον κύριο Μούρεσεν, για την παρουσία του. Μας έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση της έκθεσής του και ε, ήταν πολύ ευχάριστα για μας τα λόγια του ε, γιατί φαίνεται ότι όπως και ο κύριος Σάν είναι έτοιμος να προσπίσει τα συμφέροντα των γεωργών. Κύριε Μουρεσάν, αυτό που μας ε, ανησυχεί είναι να μην αποδυναμωθεί ο, ο γεωργικός Θέλουμε να παραμείνει ισχυρό. Και αυτό που με προβληματίζει, εδώ είμαι κύριε Μούρεσαν, εδώ στο Προεδρείο, γιατί με ψάχνατε βλέπω στην αίθουσα, αυτό που με προβληματίζει από την πρόταση των προπολογισμών είναι ότι επιτρέπεται για πρώτη φορά η ε, μεταφορά κονδυλίων από ένα τομέα σε άλλο αν το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή με τον ίδιο προϋπολογισμό θέλουμε να επιλύσουμε πολύ περισσότερες κρίσεις και αυτό ε, το πρόβλημα έχουμε και στην Επιτροπή Γεωργία όπως είπαν οι συνάδελφοι. Δεν θα πρέπει να ε, μεταφέρουμε από την Γεωργία κονδύλια σε άλλους τομείς. Και η μεταφορά ε, κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία προς άλλα ταμεία με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Δεν θα θέλαμε ε, από το γεωργικό ταμείο να μεταφερθούν κονδύλια σε άλλα ταμεία. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοια μεταφορά κονδύλιων, γιατί ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, την προσφυγική, την τρομοκρατία, να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι με το γεωργικό προϋπολογισμό. Η κοινή γεωργική πολιτική χρειάζεται ακέραιο το γεωργικό προϋπολογισμό. Και ο γεωρικό Κλάδο εξαρτάται τα μάλα από τον κοινοτικό προπολογισμό. γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τον περικόψουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σάνι και τον συνάδελφο Μούρεσαν και για την παρουσία αλλά και για την ευαισθησία που έδειξε για τον τομέα μα, Ένα τομέα ο οποίο προφανώ πρέπει να διατηρήσει υψηλή την επαγρύπνηση Ω προ το επίπεδο των προπολογισμών που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που μα περιμένουν την πρόκληση τη κλιματική αλλαγή, τη παγκοσμιοποίηση των αγορών, την πρόκληση τη σχετική με, την, ε, με το δημογραφικό, με την αναλλαγή, την ε, ποιότητα και την αηφορία των προϊόντων. Σημασία νομίζω έχει ιδιαίτερα να υπενθυμίσουμε και την ε, πρόκληση που ανέφεραν και άλλοι συναδελφοί νωρίτερα, την πτυτικότητα των τιμών Χρειάζεται λοιπόν ταχύτερη αντίδραση, πιο αποτελεσματική αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε τον αμυντικό αντίκτυπο στα έσοδα των γεωργών. Χρειάζονται δημοσιονομικοί πόροι, πρόσθετοι πόροι στον προπολογισμό του 2018 για τα γαλοκτομικά, για τα οπορολαχανικά, για τον τομέα του χείριου κρέατος για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης και του ρωσικού εμπάργου. Ιδιαίτερα όμω πρέπει να υπαγρυπνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στον φυτογειονομικό και κτηνιατρικό τομέα. 20 εκατομμύρια ευρώ μόνο προβλέπονται. Δεν μπορεί να αρκέσουν αυτά για να αντιμετωπίσουν όλο και ενισχυόμενο αριθμό ε, επιδημιών και επιζώτιων, ε, γρήπη των πτηνών και άλλα. Και βέβαια το πρόβλημα της ξυλέλα που έχει πτήσει, πλήξη της ε, ελιές, τάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση προς τον κύριο Μουρεσάν. Η Κομισιόν είπε πως ε, θα πρέπει να δούμε τα μέτρα της αγοράς ε, για τα προκυπευτικά. Πρέπει όμως να το δούμε και για τον τομέα του γάλακτος. Παραδείγματος χάρη στην Φιλανδία οι τιμές έμειναν πίσω σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών στην υπόλοιπη Ένωση και αυτό έχει οδηγήσει σε δυσκολίες και σε άλλες χώρες ε, έχουν υπάρξει εξελίξεις, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις σε σχέση με την ζήτηση. Εμείς υποφέρουμε ιδιαίτερα από το ρωσικό εμπάργο που ήταν ε, μεγάλος ο πελάτης μας και πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν αυτά υπόψη και να κινηθούμε γέρος. Θα μείνουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μουρεσάν, μιλήσατε για μια σταθερή βιώσιμη βάση των οικονομικών, μια πολύ καλή φιλοδοξία. Εντάξει, ίσως να μην ήταν τέλεια τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ε, λεφτά τουλάχιστον ε, υπήρχαν ε, και όταν μιλάτε για ίδιους πόρους, εντάξει λέτε ότι δεν θα κοστίσει περισσότερο στα κράτη-μέλη. Ε, πολλοί κόσμος δεν θα το πιστέψει, δεν φταίτε εσείς βεβαίως, αλλά φοβούμε ότι θα καταλήξετε με κάποιες ακούσιες συνέπειες. Δηλαδή, σε μια προσπάθεια να έχουμε σταθερά βιώσιμα οικονομικά, αποθούμε τον κόσμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι ίδιοι οι πόροι για εμένα χτυπάνε καμπανάκια σημαίνει τελικά μια πλήρη δημοσιονομική ένωση, ε, κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Πιστεύω στη συνεργασία εδώ με τους συναδέλφους, αλλά ε, θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίζουμε εμείς τους προπολογισμού μας και να τους διαμορφώνουμε άμεσα. Νομίζω λοιπόν πως αυτό το προτείνεται είναι λάθος, γιατί θα καταλήξουμε με μια κατάσταση ασταθή και μη βιώσιμη, ε, η οποία θα απομακρύνει τον κόσμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να παραμένουμε στο βορρά. Ο κύριος Άγνιο. Uh, Ευχαριστώ. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής στο μέλλον και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε κύριε Μουρεσάν. Ε, μιλήσατε για το τι θα γίνει μακροπρόθεσμα. Δεν αναφέρατε τα νούμερα, αλλά ο Βρετανός φορολογούμενος δίνει 6 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο και οι Βρετανοί οι γεωργοί λαμβάνουν 3 δισεκατομμύρια λίρες ε, στην κοινή γεωργική πολιτική. Τα υπόλοιπα 3 δις πήγαιναν στην υπόλοιπη Ένωση. Όταν φύγει η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλύψει αυτό το κοινό. Είτε θα παίρνουν λιγότερα λεφτά οι αγρότες ή οι πολίτες των άλλων πολιτών θα πληρώνουν περισσότερες φορές. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Ο κύριος Μορεσάν πρότεινε του ίδιου πόρου. Αυτό σημαίνει άμεση φορολογία των πολιτών από την Ένωση. Και εντάξει είναι και αυτός ένας τρόπος. Φεύγει έτσι η διακριτική ευχαίρεια από τα κράτη-μέλη. Αλλά το συγκεκριμένο μου ερώτημα είναι εάν αυτό θα απαιτήσει αλλαγή της συνθήκης, γιατί είναι σοβαρή αλλαγή. Ευχαριστώ κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φοβόμουν ότι όντω θα χρειαστεί να λάβω το λόγο αμέσω μετά τον κύριο Άγνιο. Ξεκινώντα, επισημαίνω ότι δεν σκόπευα να λάβω το λόγο. Γιατί ομολογώ ότι δεν είμαι ειδικό στα δημοσιονομικά. Αλλά θα πρέπει να, να ομολογήσουμε όλοι ότι ο ο Γεωργικός Προπολογισμό έχει πολύ μεγάλο μερίδιο από τον Ευρωπαϊκό. Ανέφερε ο κύριος ε, Μουρεσάν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Είχαμε το γαλακτοκομικό, την γρήπη των πτηνών πέρσι. Έχουμε ακόμη την ε, κρίση με το εμπάργο το ρωσικό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι είδους κρίση μπορεί να προκύψει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Μπορεί να προκύψει μια μικρή, μια μέτρια ή μια τεράστια κρίση. Ο λόγος όμως προκύπτουν αυτές οι κρίσεις είναι ότι είναι πολύ βραδία η ανταπόκριση. Και εδώ ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Σαντέρ όταν λέει ότι θα μπορούσαν με ταχύτερη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτές οι κρίσεις να μην έχουν τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Και συνέπειες και το είδαμε αυτό με την κρίση στο γαλακτοκομικό αλλά και σε άλλους τομείς. Άρα χρειάζεται ταχύτερη ανταπόκριση και πιστεύω ότι αυτό προσπαθεί να παράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω θέσει διαφορετικέ βέβαια με τον κύριο Άγνιου, αλλά δεν μπορώ παρά να ομολογήσω ότι επισημαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα για τον προπολογισμό με, με τη ρένα εξελίξη η πολιτική, όταν δηλαδή εν τέλει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Είπε ο κύριο Άγνιου ότι πρόκειται για 6 δι. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα καταλαβαίνω πολύ τα οικονομικά αυτά. Αλλά τι συνέπειε θα έχει όσο προχωρήσει αυτή η υπόθεση, γιατί σου χρειαστεί να ξανακαθίσει στο τραπέζι να συζητήσουν ε, η ευρωπαϊκή πλευρά με το Ηνωμένο Βασίλειο και το κόμμα του κυρίου Άγνιου μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να δώσει περισσότερα χρήματα για τους γεωργούς από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω κανένα γεωργό στην Ευρώπη να βρεθεί σε θέση δυσμενέστερη επειδή αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα πρέπει η Επιτροπή των Προπολογισμών να το κοιτάξει αυτό σαν πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την αλληλουχία αυτών των παρεμβάσεων παρόλο που ήταν τυχαία αλλά τελικά ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ τους κυρίους Σάνι και Μουρεσάν και να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκολσον για το γνήσιο ενδιαφέρον του για τους γεωργούς της Ευρώπης γιατί είναι μέλος ε, του, από το Ηνωμένο Βασίλειο και μας ενδιαφέρουν οι δικές ανησυχίες για το θέμα αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι σοφός άνθρωπος ο κύριος Νίκολσον. Δεν το λέω συχνά, αλλά είναι πολύ σοφός άνθρωπος και έχει μακρά πείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ε, και θα πρέπει να εξεράσουμε την εκτίμησή μας για τον τρόπο τον οποίο ρίμισε για τους Γιώργους. Αλλά και εγώ ενδιαφέρομαι ε, για του ε, γεωργού του Ηνωμένου Βασιλείου, όπω ο κύριο ενδιαφέρεται για του υπόλοιπου Ευρωπαίου γεωργού, γιατί είναι μικρή φωνή του σε μια μεγάλη χώρα. Ε, και στην ε, προεκλογική εκστρατεία που ε, θα παρακολουθήσουμε, θα θέλαμε να δούμε ποια θα, ποια θα είναι τα σχέδια για την γεωργική πολιτική και την πολιτική των τροφίμων του Ηνωμένου Βασίλειου. Θα έχει ενδιαφέρον και για εμά. Και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2018, γενικώ το πρόβλημα που έχουμε με του προπολογισμού είναι έχουμε ένα πάγιο τμήμα που προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε σε ένα κινητό ε, τμήμα που αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Ε, εκτίμησα ιδιαίτερα από την παρουσίασή σας το πραγματικό ενδιαφέρον και τη γνώση σας ε, για τη γεωργία. Και ελπίζω τουλάχιστον μερικές δεσμεύσεις να τις στηρίσετε, γιατί θέλουμε μεγαλύτερη ε, δέσμευση των μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τη Γεωργία. Και αν θέλουμε να αναπτύξουμε την κοινή μας γεωργική πολιτική σήμερα, θα πρέπει να δούμε τους στόχους μας και να εξασφαλίσουμε περισσότερα κονδύλια για να τους υλοποιήσουμε, ιδιαίτερα τα δημόσια αγαθά και δεδομένου της τιμή ε, των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Ε, ναι, διαχείριση των κρίσεων στη Γεωργία. Τι ωραία φράση. να, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ανάπτυξη μέσω της κρίσης, ε, για την αξιοποίηση των ευκαιριών που μας δίνει η κρίση, γιατί και αυτό ίσως έχει σημασία. Ο γραμματέας κανόνισε την ακολουθία των παρεμβάσεων. Δεν έγινε καμία ε, δεν ήταν καθόλου προσχεδιασμένη. Αλλά πραγματικά ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η συνέχεια, η σειρά των ομιλιών. Μπογκόβιτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή η αλουχία των παρεμβάσεων. Ε, Βεβαίω και αντιλαμβάνομαι ότι το Brexit θα προξενήσει κεφαλό και σε αυτούς που αποχωρούν και σε αυτούς που μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 μάλλον δεν θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις από αυτό, αλλά και θα ήθελα να προσθέσω και να επαναλάβω ότι είναι πολλές οι κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο, ειδικότερα ο γεωργικός Τοπέα. Ο παγετός, παραδείγματι, για δεύτερη χρονιά η Σλοβενία έχει αντιμετωπίσει ε, ολοκληρωτική απώλεια παραγωγής Ε, εγώ με τρία εκτάρια μόνο που είχα κανονικά 150 τόνους παραγωγή μήλων αχλαδιών, τώρα μπορώ να περιμένω 10 με 15 το πολύ πολύ. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε και πέραν της ασφάλισης αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί είναι χαμηλές επιδοτήσεις στη χώρα μου. Και βέβαια συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια οι Γεωργοί, αλλά για να μιλήσω και για τα εκκρεμή ζητήματα, η Σλοβενία υιοθέτησε πέρσι έναν ειδικό νόμο, ο οποίο όμω δεν καλύπτει την απώλεια εισοδήματος τη προηγούμενη χρονιά για τους γεωργού και άρα μένουν οι γεωργοί για δεύτερη χρονιά χωρί εισόδημα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε επαρκή κονδύλια και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά αλλά και των λοιπόν κινδύνων. Χρειάζεται μια πιο αποφασιστική πολιτική για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγής. Και αυτό ταχύτατα. Ιδάλλως η παραγωγή ε, γενικά τροφίμων ε, ο πορολαχανικών, ή, ε, κλίμα, η αμπελιού θα καταστραφούν. Είναι πρόβλημα οι κλιματικέ αλλαγέ και δύσκολο θα τι αντιμετωπίσουμε γρήγορα. Θα ήθελα να καλωσορίσω α, ε, τους ε, καλεσμένους του κυρίου Έρντος από την Ουγγαρία. Καλώς ήρθατε. Πρόκειται για εκπροσώπου ε, οργανώσεων παραγωγών. Μένουμε στο Νότο τώρα, η κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων των φορολογουμένων και να προλαμβάνουμε κάπως τα προβλήματα, να είμαστε πιο διορατικοί για να προασπίσουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των πολιτών μας και ιδιαίτερα των γεωργών. Η κρίση που έπληξε, η κρίση που έπληξαν τον γεωργικό τομέα ήταν πολλές και γι' αυτό χρειαζόμαστε ιδιαίτερο τμήμα του προπολογισμού για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Και αυτά τα κονδύλια δεν θα πρέπει να προέρχονται από το γεωργικό προπολογισμό. Το ρωσικό εμπάργκο έπληξε τον γαλακτοκομικό τομέα και τον τομέα των απορακυπευτικών. Επίση, μεταξύ καταργήθηκαν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσει. Είχαμε τι θεομηνίες και πέρυσι και φέτος. Και εμεί φέτος ακόμη μετράμε τι ζημιέ από τι θεομηνίες. Επιπλέον έχουμε τεράστια στάθεια στις αγορές και στις τιμές. Δεν μπορούν από μόνοι τους οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις κρίσεις. Αλλά ούτε και τα κράτη-μέλη έχουν αρκετά κονδύλια για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απροσδόκητες κρίσεις. Και οι γεωργοί περιμένουν πολλά από εμά, ιδιαίτερα από τους Ευρωβουλευτές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τους δώσουμε την κατάλληλη απάντηση, γιατί έχουμε 12 εκατομμύρια γεωργού που με μεγάλη δυσκολία προσπαθούν να εξασφαλίσουν παραγωγή τροφίμων για τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω ότι ε, χρήζουν τη ε, ε, υποστήριξή μα και τη υποστήριξη των δικαιωμάτων του. Παραμένουμε και πάλι στο Νότο, κύριο Δεκάστρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μερικά δευτερόλεπτα μόνο θα σας απασχολήσω. Θέλω να ευχαριστώ τον συνάδελφο Τιμποσάνη και τον κύριο Μουρεσάν για τι τοποθετήσει και την ειλικρίνεια που επέδειξε σήμερα για τη γεωργική πολιτική. Πολλοί συναδελφοί υπενθύμησαν ότι ζούμε σε μια περίοδο αβεβαιότητα, σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι και οι κρίσεις εναλλάσσονται και θα πρέπει να φροντίσουμε να εξυγχρονίσουμε αυτή τη γεωργική πολιτική της Ευρώπης ώστε να την καταστήσουμε πιο ε, κατάλληλη για να στηρίξει τους ε, γεωργούς και να τους αντιβοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Κάτι μικρό ήδη μπορούμε να πράξουμε αύριο με την έγκριση του κανονισμού Omnibus που θα σημάνει κάποια βήματα πρόοδου στη διαχείριση ακριβώς των κινδύνων. Σύμφωνα και εγώ με την κυρία Μαγκίνες υπογραμμίζοντας πόσο σοφός είναι ο Τζιμ Νίκολσον και θέλω να υπενθυμίσω στον συνάδελφο Άγνιου ότι το 1984 πληρώνουμε το Βρετανικό rebate, ε, την έκπτωση, επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικού μέρου των πόρων της συνεισφορά του. Άρα λοιπόν ε, αυτή η διαφορά που μπορεί να σας φέρετε ότι είναι εις βάρος του Βρετανικού λαού είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι επισημαίνετε εσείς. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier... Ο κύριος Δαντάν, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ τους ε, δύο συγητές, τον ε, κύριο Σάμπορ και τον ε, Γενικό Εισηγητή και θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν ορίστηκαν τα πολύτιμη νομικά πλαίσια της τρέχουσας περίοδου. Όλες οι ενδείξεις έδειχναν ανάπτυξη, ανάπτυξη της κατανάλωσης αλλά και της ζήτησης ω εκ τούτου και των τιμών. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ορισμένοι θεωρούσαν ότι ήταν έως και περιττό να προβλεφθούν τότε το 2013 εργαλεία διαχείρισης της κρίσης. Άλλαξαν όμως ταχύτατα τα πράγματα, πολύ ε, έντονα και βλέπουμε μια αλλαγή κατάσταση σε βαθμό που από το 2014 η μία κρίση ε, ακολουθεί την άλλη, είτε πρόκειται για ε, κρίση κοινωνική, δεοντολογική, ηθική, κλιματική, οικονομική. Μπορούμε να απαντήσουμε βέβαια αποτελεσματικά μόνο στην κλιματική και οικονομική κρίση και ως εκ τούτου οτιδήποτε και αν προκύπτει από τους άλλους τομείς ως αιτήματα, Φερρυπίν, το μεταναστευτικό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, παραμένει μεγάλη ανάγκη για μια ισχυρή γεωργική πολιτική με προπολογισμό βέβαια εισάξιο. Ευχαριστώ πολύ. Ας δούμε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να πει. Η Διευθυντρία έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος κι εγώ. Να επαναλάβω ότι η Κομισιόν είναι διατεθειμένη σε περίπτωση κρίσης να παρέμβει. Το 2015, 2016 και 2017 έχουμε υποβάλει ένα πακέτο 1,7 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τις ε, συνέπειες της ρωσικής κρίση σε μεγάλο ποσό νομίζω και αυτό έγινε δυνατόν χάρη στο ότι και το Κοινοβούλιο κατέληξε γρήγορα σε μια έκθεση γιατί όπως είπαν πολλοί ε, βουλευτές όταν υπάρχει κρίση σημασία έχει να αντιδρά κανείς γρήγορα και αυτό ε, κατέστη δυνατόν χάρη στην δική σας στήριξη. Μπορώ να σας πω ήδη σήμερα ότι το 2018 για το σχέδιο προπολογισμού θα υπάρξει συνέχεια κάποιων μέτρων για οπωροκυπευτικά γιατί όπως είπατε οι δυσκολίες συνεχίζονται και υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε τους αγρότες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κρίση. Ίσως ένα συγκεκριμένο θέμα να αναφέρω που ανέφερε ο εισηγητής να υπάρχει αρκετό περιθώριο το 2018 για την Γεωργία. Ναι, βεβαίω αυτή είναι η πρόθεση της Κομισιόν. Αλλά γνωρίζετε όλοι πως όσον αφορά τις ε, πιστώσεις ε, πληρωμών το 2018 και τα επόμενα έτη θα είναι πιο δύσκολα γιατί θα υπάρχει μια αύξηση στο, ε, στα διαρθρωτικά ταμεία κάτι το οποίο θα μειώσει το περιθώριο λιγμών σε πιστώσεις πληρωμών. Και ξέρετε ότι αυτό θα επηρεάσει την ε, αγροτική ανάπτυξη. Όμως θεωρώ ότι τα περισσότερα από τα σχολεία σας θα υιοθετηθούν και θα το δείτε αυτό στο τέλος Μαΐου όταν θα παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού η Κομισιόν. Νομίζω πως υπάρχει λοιπόν μια συναντήληψη εδώ των δύο θεσμικών οργάνων για τον προϋπολογισμό του 2018. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα ακούσω τώρα το, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μουρεσάν, τον εισηγητή. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, γιατί μίλησα πολύ στην αρχή. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τους συναδέλφους που μου έδωσαν μια καλύτερη εικόνα του που βρισκόμαστε, ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, του τομέα της Γεωργίας ε, το έτος που έρχεται. Ο Άλμπερτ Ντές μας είπε το πόσα καταφέραμε να επιτύχουμε μέσω των δαπανών στην Γεωργία και γι' αυτό νομίζω πρέπει να υπερασπιστούμε μαζί τις δαπάνες στον τομέα της γεωργίας ως επενδύσεις στην ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στις θέσεις εργασίας όπως ανέφερε και η συνάδελφος θέσεις εργασίας στην υπαίθρο σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις συχνά και βεβαίω ε, στην Υπεθρό όπω όπως είπε και η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία Γκαρθία Α, ναι, βρούμε κάποιες νέες προτεραιότητες, το είπα και εγώ στην αρχή, νέες προτεραιότητες που δεν υπολογίζαμε στην αρχή του πολιετού δημοσιονομικού προγράμματος. Αυτό πρέπει να γίνει με φρέσκα κονδύλια και ε, καινούργια δηλαδή α, ε, α, ε, κονδύλια και όχι εις βάρος της Και βεβαίω ο κύριος Σάγκιο ανέφερε την ε, σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου ότι συνεισφέρει δηλαδή στον προϋπολογισμό ωφελείται κιόλα, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος δικαιώχος π.χ. ο προϋπολογισμός ε, έρευνας και καινοτομίας ε, λόγω των Βρετανικών Πανεπιστημίων τα οποία είναι κορυφαία και ωφελούνται πολύ περισσότερο και ήταν πράγματι ε, κάτι το ε, πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να τα δούμε συνολικά για να είμαστε ειλικρινεί με τους πολίτες μας. Συνολικά λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να παραμένουμε σε επαφή ειδικά αφού παρουσιάσει ένα σχέδιο προπολογισμού η Κομισιόν και θα έχουμε και νούμερα για αυτά τα οποία γράφει ο Τίμπορ στην γνωμοδότησή του. Όταν λοιπόν έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς από την Κομισιόν, θα αναμένω και την άποψη της Επιτροπής σας για την πρόταση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ και καλή συνεδρία Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Ευρωβουλευτά. Ο αριθμός των επένων, άντε καλά μιλάτε ίσως αργότερα, ο κύριος Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους γιατί ήταν ο διάλογός μας ένας από τους πιο καρποφόρους ε, διαλόγους στην Επιτροπή γιατί έχουμε καθορίσει πολύ καλά τις προτεραιότητες και το που δίνουμε έμφαση και νομίζω ότι ε, όλα αυτά θα αποτελέσουν πολύ καλή βάση για συνεννόηση της Επιτροπής Γεωργίας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και να πω και δύο λόγια ακόμη. Φαίνεται να μιλάμε για χρήματα, μια και ασχολούμαστε με τον προπολογισμό, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι κυρίως πολιτικό. Και το θέμα που θα πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε και προς τον έξω κόσμο, προς το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι μία από τις ε, ουσιώδεις βασικότερες αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο ένας απλός κλάδος, δεν είναι μια τομεακή πολιτική. Αγγίζει το πύρι, τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα την αναπτύξουμε. Και χαίρομαι που πολλοί συνάδελφοι τόνισαν ιδιαίτερα τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Γιατί αυτά είναι εργαστήρια που σχεδιάζουμε το μέλλον. Και σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε τον τομέα αυτό. Και αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι μόνο η διασφάλιση ε, του γεωργικού τομέα που θα πρέπει να γίνει, αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και προς τους συμπολίτες μας θα πρέπει να σκεφτούμε και μια αναζωογόνηση της υπαίθρου, όχι μόνο μια διατήρηση και διασφάλιση του γεωργικού κλάδου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε λάβει τόσες πολλές παρατηρήσεις, τόσα πολλά σχόλια, τόσα πολλά εγκόμια και πένους που πραγματικά σας τροφοδοτούν για περαιτέρω πολύ εντατική εργασία. Και αυτό σας ευχόμαστε. 29 και 30 Μαΐου θα εγκρίνουμε την γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα εγκρίνει τη δική της έκθεση 19 και 20 Ιουνίου, ενώ η έγκριση στην Ολομέλεια θα γίνει στην πρώτη Ολομέλεια του Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και συνεχίζοντας την πρόταση του κύριου Ντές, θα ήθελα να σας ξανακαλέσω στην Επιτροπή μας για συνέχιση των συζητήσεων. τώρα στο επόμενο θέμα, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία τη Χιλή για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Εμεί θα συντάξουμε γνωμοδότηση για την οποία αρμόδια είναι η κυρία Γκιλέρα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτριά μα. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ε, συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα αναγνωρίσει αμοιβαία την ισοδυναμία των κανόνων βιολογικής παραγωγής και των συστημάτων ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Χιλή. Η συμφωνία αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο Φαντάζομαι ότι έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό, γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής, η Γενική Συμφωνία, η Γενική Συμφωνία Εμπορίου με τη Χιλή, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Η συγκεκριμένη συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια των συμφωνιών νέας γενιάς, όπως τις αποκαλούμε. Επαναλαμβάνω, σχετική συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, ε, έχουν γίνει δεκτά κάποια προϊόντα από τη Χιλή, όχι όλα. Και λόγω ελέγχων που έγιναν, φαντάζομαι ε, έχουν αποκλειστεί ε, τα λοιπάσματα, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας ε, και το κρέας. Προς το παρόν τουλάχιστον έχουν αποκλειστεί αυτά τα προϊόντα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή. Η συγκεκριμένη συμφωνία ε, που αφορά βιολογικά προϊόντα έχει δύο ζητήματα. Πρώτη φορά καταρχήν συνάπτουμε έκθεση σε ε, συμφωνία τέτοιου επίπεδου. Και η πιο σημαντική καινοτομία της συμφωνίας αυτής είναι ότι ακριβώς και πρώτη φορά αναγνωρίζονται σε μία συμφωνία οι ισοδυναμίες. ισοδυναμίες των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω ακούσει, ενώ έχουμε συμφωνίες με 14 χώρες, καμία από αυτές ε, δεν έχει την ισχύ συνθήκης. Είναι διμερούς χαρακτήρα. Οπότε, η καινοτομία έγκυται όχι στο ότι έχουμε αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μια άλλη χώρα, γιατί αναγνωρίζουμε βιολογικά προϊόντα και από όλε 14 χώρε. Η καινοτομία έγκυται στο ότι για πρώτη φορά η συμφωνία αυτή έχει το χαρακτήρα συνθήκη. Αναγνωρίζεται σε συνθήκη. Και μάλιστα για πρώτη φορά σε μια συνθήκη έχουμε αναγνώριση τη ισοδυναμία των κανόνων παραγωγή και συστημάτων ελέγχου. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από την ε, Επιτροπή Γεωργίας ότι παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία και έχει υπογραφεί έχουμε τώρα τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, αυτό προβλέπει η διαδικασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θα ήθελα πάντως να πω ότι κατά τη γνώμη μου οι διαδικασίες αυτές δεν συνάδουν με, την, ε, με τον δέοντα σεβασμό που οφείλει η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί μιλούμε για μια γνωμοδότηση που αφορά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής, η συμφωνία όμως που ήδη έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί. Οπότε τι γνωμοδότηση δίνουμε κατόπιν εορτής. Ε, άλλωστε αρμόδια κατ' ουσίαν είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εμείς απλή γνωμοδότηση δίνουμε. Και αυτή είναι η συνηθισμένη διαδικασία. Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά δεν μπορώ να μην εκφράσω την αντίρρησή μου, γιατί θεωρώ ότι δεν γίνεται σεβασμό, σεβαστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή, παρόλο που είναι η συνήθις διαδικασία. Έχουμε μία συμφωνία για την οποία μπορούμε απλώς να πούμε ναι ή όχι. Δεν έχουμε δυνατότητα τροποποίησης. Στη γνωμοδότησή μου αναφέρθηκα σε κάποια σημεία. Καταρχήν αναθεωρείται ο κανονισμός για τη βιολογική γεωργία. Οπότε η συμφωνία αυτή που έχει προηγηθεί της αναθεώρησης του κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί κάποια στιγμή με τον αναθεωρημένο προπολογισμό. Και αυτό ζητώ στη γνωμοδότησή μου. Ότι μια και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να συνάδει με τη νέα νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή όταν εγκριθεί. Άλλο θέμα είναι το θέμα των συνεπειών, του αντικτύπου. Θα πρέπει ο αντίκτυπος να λαμβάνεται υπόψη κατά την υπογραφή μιας συμφωνίας με τρίτη χώρα. Και όχι μόνο ε, οι συνέπειες εκ των υστέρων, αλλά και εκ των προτέρων. Δηλαδή θα πρέπει εκ των προτέρων να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες συγκεκριμένων προϊόντων στις χώρες αυτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε μόνο για βιολογικά προϊόντα. Και το αίτημα για βιολογικά προϊόντα, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά την παραγωγή ε, βιολογικών προϊόντων. Είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε τέτοια προϊόντα και αυτό ισχύει γιατί και από τη Χιλή εισάγουμε βιολογικά προϊόντα. Θα αυξηθεί το σχετικό εμπόριο 5% ετησίως και μάλιστα αυτό συνέβη και την τελευταία δεκαετία, γιατί θα αυξηθεί η παραγωγή και στο μέλλον, αλλά υπάρχει και αύξηση τη ζήτηση, ακόμη και τη εσωτερική ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί η κοινοτική παραγωγή βιολογικών προϊόντων για να καλύψει την ζήτηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εισαγωγή. Εγώ ε, συνέταξα την έκθεση την γνωμοδότησή μου μάλλον προκειμένου να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Άλλωστε μόνο δικαιούμαστε να πούμε ναι ή όχι για τη συμφωνία. Σας εξέφρασα τις αμφιβολίες μου. Το μόνο που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί τελικά είναι το ναι ή όχι εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Αύριο θα γίνει η συζήτηση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Και επαναλαμβάνω, η, έκθεση έχει ήδη, η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί και επαναλαμβανω η εκθεση η συμφωνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Χίλη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τη Μαρία Άγγελος που είναι εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, για ποιο λόγο αποφασίσετε να διαχωρίσετε τα βιολογικά προϊόντα και να συνάψετε ξεχωριστή συμφωνία στο, στο περιθώριο της συμφωνίας γενικού εμπορίου που έχετε με τη Χιλή. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ανάγκασαν να διαχωρίσετε τα βιολογικά προϊόντα. Για ποιους λόγους τα διαχωρίσατε. Επίσης, κάτι που με ρώτησαν οικολογικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτή η ισοδυναμία της, των κανόνων που μέχρι στιγμής γινόταν σε διοικητικό επίπεδο. Τι συνέπειες θα έχει εφόσον κατοχυρώνεται σε συνθήκη θέλουμε να ενημερωθούμε για τις συνέπειες που θα έχει η αναγνώριση της ισοδυναμίας των κανόνων τώρα που η ισοδυναμία αυτή αναγνωρίζεται σε μια συνθήκη και όχι απλώς διοικητικά. Επαναλαμβάνω, δεν μου άρεσε ούτε ο τρόπος ε, ε, διεξαγωγής των συζητήσεων, ούτε η συνήθις διαδικασία που φέρνει το Κοινοβούλιο να αποφαίνεται κατόπιν εορτής μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Αυτές τις ε, κριτικές βέβαια τις έχετε ξανακούσει γιατί στυλιτεύουμε αυτή την αδιαφάνεια και την ε, πολύ εκ των υστέρων ε, διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μας ενδιαφέρει να δίνουμε τη γνώμη μας που θα είναι απλώς ένα ναι ή ένα όχι και μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Θα θέλουμε στο μέλλον να τροποποιηθούν οι διαδικασίες. Και σας είπα ποια είναι η γνώμη μου για τη γνωμοδότηση. Παρ' όλα αυτά είμαι υπέρ της συμφωνίας με τη Χιλή με τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες που εξέφρασα και κυρίως ε, μεγάλη επιφύλαξη για το θέμα των, της ισοδυναμίας και ρώτησα τι αντίκτυπο θα έχει συνθήκη, το καθεστώς της συνθήκης στο θέμα αυτό. Μάλιστα, παίρναμε στη συζήτηση. 1,5 λεπτό στον καθένα. Ο κύριος Στάκουλα πρώτος, 1,5 λεπτό επαναλαμβάνω. Thank you, Chair, dear colleagues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λίγα λόγια. Όπως ξέρετε, είμαι μέλος και στην Επιτροπή Εμπορίου Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία για βιολογικά προϊόντα που θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς φτάνεται συνεχώς η παραγωγή αυτού του κλάδου εκτιμάται πως ο κλάδος αναπτύσσεται την τελευταία δεκαετία συνεχώς. Η προτινόμενη συμφωνία δεν έχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Η χιλή δεν έχει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα. Ε, είναι ο λιγότερο προβληματικός εταίρος στην ε, Νότια Αμερική. να Έχουμε τις ίδιες αξίες. Κάτι πρέπει να πούμε ότι ε, η προτινόμενη συμφωνία πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό βιολογικής παραγωγής και την τελευταία του ενημέρωση. Ένα άλλο σημείο που αναφέρει η γνωμοδότηση ήταν η αίτηση για αξιολόγηση αντικτύπου, την οποία στηρίζω πλήρως καθώς πρόκειται για την πρώτη τέτοια συμφωνία και πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιδιώκεται μια ακόμη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η οποία θα επιδεινώσει συνθήκες ανταγωνισμού για τους παραγωγούς, τους Γάλλους αλλά και τους Ευρωπαίους έτσι λοιπόν τα κρασιά, τα επιτραπέζια στα φίλια θα πλήξουν, θα έρθουν από την χειλή για να πλήξουν τους παραγωγούς μας. Και πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα τα παράγουμε με άλλους όρους εδώ. Είναι ανόητο λοιπόν το σύστημα και επιβαρύνει πολύ έναν ίδιο θέμα του ανταγωνισμού. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Τι μας αποφέρει αυτή η συμφωνία για τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Δεύτερον, σε τι τιμές θα πολλούνται τα προϊόντα αυτά. Και άλλη μια ερώτηση για τα βιολογικά προϊόντα που έχουν ξεκινήσει για διάφορους λόγους και για να ε, τρώμε πιο υγιεινές τροφές αλλά και για να ευνοείται ε, μια διαδρομή σύντομη κατά το δυνατόν του προϊόντος μέχρι το τραπέζι του καταναλωτή. Σε τι εξυπηρετεί λοιπόν να έρχεται από, το, από τη χιλή, από τόσα χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα και να επιβαρύνει και το, η κλιματική αλλαγή με διοξείδιο του άνθρακα και αέριο του θερμοκηπίου, όταν βιολογικό σημαίνει ότι μειώνουμε όσο δυνατόν την απόσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Σουλάνακαν. Όταν πρωτοδιάβασα ότι υπήρχε το θέμα αυτό στην εμερική διάταξη, έδειψα τα μάτια μου, το ξαναδιάβασα και το διάβασα. γιατί δεν ευχαριστώ και νόημα. Είναι σαν να μας λέτε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα βραβείο σοκολάτας μέσα σε μία τσαγέρα με σοκολάτα. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα, θα έρχονται από τη χιλή. Κάποιος ζήτησε εξηγήσει. Καταρχάς υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση για τέτοια προϊόντα, ε, ας τα παράγουμε εδώ. Όταν, κάτι, όταν ένα προϊόν κυκλοφορεί από την άλλη άκρη του κόσμου μέχρι εδώ, πώς θα πάρει το, την ετικέτα του βιολογικού. Δεν μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ή, πάση περιπτώσει, σε ποιον πλανήτη ζούμε. Ευχαριστώ κύριε Στενανό. Όχι, ο κύριος Oui. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ θα υιοθετήσω τις ε, προτάσεις της Κλέρα Αγγουιλέρα. Είναι εύστοχα τα ζητήματα που θέτει, τα υιοθετούμε. Και βεβαίως υπάρχει η στιγμή αποτύπωση της βιολογικής παραγωγής, αλλά και η διαδρομή. Αυτή η στιγμή είναι σε επεξεργασία ο σχετικός κανονισμός και θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα, όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε. Έτσι λοιπόν... Τώρα μας λέτε να πούμε το ναι ή το όχι, αλλά ή μη τι άλλο. Ας εμπνευστούμε από τους νέους κανόνες που όπου να είναι θα ε, θεσπιστούν. Είναι λίγο παράξενη αυτή η κατάσταση να προχωρούμε σε έγκριση ενός κανονισμού και από την άλλη να μας δείτε η έγκριση μιας ε, συμφωνίας που έχει ε, συναυθεί από διαφορετικές συνθήκες. Και η απόσταση βεβαίως. Υπάρχουν πολλά αισθήματα λοιπόν που πρέπει να ρυθμιστούν στα βιολογικά παραδείγματα τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν νομοθεσία και ξέρω ότι βεβαίως ε, δίνουμε απάντηση μέσα από συμφωνίες συμμόρφωσης. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα σύστημα συμμόρφωσης για τα προϊόντα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και το σύστημα της ισοδυναμίας, τη ισοτιμία προϊόντων για χώρε που έχουν τέτοια συστήματα όπω η Χιλή. Πρέπει λοιπόν να τα κοιτάξουμε προσοχή. Και επίσης όπως είπα, η χρονική στιγμή που θα εξετάσουμε έχει να κάνει και με την απόσταση που είναι πολύ μεγάλη. Και ναι, βέβαια πρέπει να ενθαρρύνουμε τον Ευρωπαίο παραγωγό σε μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το ε, ορίσουμε με διάταγμα και ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα συμβεί. Ας ενθαρρύνουμε τη βιολογική παραγωγή, την εγκύτητα, το συσχετισμό των παραγωγών και ας ρυθμίσουμε τις αγωγές και εξαγωγές όπως γίνεται μέσα από αυτή την έκθεση. Αλλά ας είμαστε προσεκτικοί. Όπως είπα, υπάρχει η στιγμιαία αποτύπωση, αλλά και η ευρύτερη θεώρηση μέσα από τις ε, γενικότερες διατάξεις και περιμένω πολύ μεγάλη όρεξη της απαντήσεις Επιτροπής. Κυρία Σάνδρα. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτριά μας, την κυρία Αγγιλέρα. Ως προς την ουσία όμως δεν συμφωνώ καθόλου με τη σύναψη της συμφωνίας αυτής με τη Χιλή. Ως εκ τούτου εγώ θα καταψηφίσω τη γνωμοδότηση. Γιατί θεωρώ ότι η βιολογική γεωργία δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας, ε, μία μέθοδος παραγωγής. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απασχόληση, τις συνθήκες των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εγκύτητα. Δεν μπορεί να είναι ένα γεωρικό μοντέλο που θα συμβάλλει στην ενεργειακή κατασπατάληση ή στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου ή στην ενίσχυση των κλιματικών αλλαγών. Η εναλλακτική λύση, όχι μόνο για τη βιολογική γεωργία, αλλά κυρίως για τη βιολογική γεωργία, ιδιαίτερα για την βιολογική γεωργία, είναι η πρόθεση της τοπικής βιολογικής παραγωγής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ε, είναι δυστυχώς υπανάπτυκτη σε πολλές ε, χώρες. Επίσης θα πρέπει να καταναλώνουμε εποχιακά προϊόντα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Το διεθνές εμπόριο, το μαζικό διεθνές εμπόριο και η μαζική κυκλοφορία βιολογικών προϊόντων ε, στον πλανήτη ή αντιβαίνει πλήρως με την ανάγκη της συμβολής του γεωργικού μοντέλου στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Κύριε κυρία Πετήρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμφωνία. Μπορούμε μόνο να την στηρίξουμε, να την απορρίψουμε, αλλά να την αξιοποιήσουμε για να διαρωτηθούμε ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη τέτοιων συμφωνιών. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πιο ισχυρός ε, στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Ε, η Χιλή θα μπορεί να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά γεωρικά προϊόντα και κρασιά μεταξύ άλλων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να ε, εξάγει τα προϊόντα της προς τη Χίλη και τα ευρωπαϊκά δηλαδή κρασιά μπορούν μεταξύ των άλλων προϊόντων να εξάγονται προς τη Χιλή. Θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε ένα δίδαγμα και να δούμε τι αποτελεσματικά μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τη βιολογική παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην χρειάζεται να προσφεύγουμε σε εισαγωγές γιατί η ζήτηση βιολογικών προϊόντων έχει αυξηθεί οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε και υπάρχει αύξηση κατά 5% των βιολογικών προϊόντων ε, ετησίως. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε την αγορά, αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε τη δική μας παραγωγή. Γι' αυτό χρειάζονται μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο γιατί στηρίζω αυτό το οποίο είπαν πολλοί συνάδελφοι ότι πρέπει να περιοριστούμε περισσότερο στην τοπική παραγωγή και ελπίζω να με στηρίξουν και αυτοί οι συνάδελφοι στο ότι πρέπει να εμποδίσουμε ε, ο Επίτροπος ε, να απαγορεύει συνεχώς ε, τις εκτάσεις προτεραιότητας για την απαγόρευση μέσων φυτοπροστασίας. Εάν γίνει αυτό θα χάσουμε αυτό το 1 εκατομμύριο τόνους και θα πρέπει να εισαχθούν αυτές οι ποσότητες από την Νότια, από Αμερική, κάτι το οποίο σημαίνει 40 εκατομμύρια τόνοι καύσιμα εκτός των άλλων. Θα πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε αυτές τις ε, προθέσεις της ε, Κομισιόν και του Επιτρόπου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπενίτα Σαράς είναι εκπρόσωπος της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Θα ήθελα να της δώσουμε το λόγο. Α, συγγνώμη. Προηγείται ο κύριο Άγνιου, συγγνώμη. Πρώτα ο κύριο Άγνιου. Ναι. Νόμιζα ότι είδατε την κάρτα μου. Δεν ε, τη σήκωσα τελευταία στιγμή. Λοιπόν, η βιολογική παραγωγή είναι κάτι το υποκειμενικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω κότες ελευθέρας βοσκής, ε, τις οποίες ταΐζω βιολογική πρωτεΐνη και παράγουν κοπριά, την οποία μου επιτρέπεται να πουλήσω ε, σε γεωργούς για... που παράγουν και εκείνοι με την σειρά τους ε, βιολογικό στάρι. Και αυτό επειδή είναι ελευθέρας βοσκής τα κοτόπουλά μου υπερισχύει του ότι τα ταΐζω γενετικά τροποιημένα τρόφιμα. Και επιτρέπεται. Οπότε αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι τα τοπικά ε, τρόφιμα είναι πιο σημαντικά από το να ε, τηρούνται οι βιολογικές αρχές. Δεν τους αρέσει το να κουβαλάνε τα τρόφιμα από την άλλη άκρη του κόσμου, όπως είπε ο κύριος Φλάναγκαν. Δεν το θεωρούν πολύ βιολογικό. Οπότε η μόνη λύση είναι οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων να απαιτούν σωστή σήμανση. Από πού ήρθε το τρόφιμο, πώς παρήχθη, με ποιους κανόνες και ποιοι κανόνες παραβιάστηκαν και έτσι να λάβουν μια απόφαση. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε όμως κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα εκπρόσωπο τη γενική Διεύθυνση Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ε, αποσαφηνίζονται καλύτερη απόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ε, με στεναχωρεί να λέει η κυρία Αγγιλέρα ότι δεν σεβόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αντίθετο Ίσα ίσα σεβόμαστε ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λαμβάνουμε υπόψη την άποψή του σε όλε τι ενέργειε μας. Και όπως είπατε και εσείς κυρία Αγγιλέρα, ακολουθήσαμε τη συνηθισμένη διαδικασία, το αναγνωρίσατε και εσείς. Δεν απομακρυνθήκαμε επουδενή από τη διαδικασία αυτή. Και μάλιστα, είχαμε δύο ευκαιρίες συνάντησης. Τον Νοέμβριο του 2015, κατά την έναρξη των συζητήσεων και πέρυσι κατά τη μονογραφή της συμφωνίας. Αν κάποια στιγμή νιώσατε ότι ε, δεν δείξαμε το δέοντα σεβασμό το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λυπάμαι, αλλά πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτή η πρόθεση ούτε και η, ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις, να πω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά μόνο τα βιολογικά προϊόντα. Είχαμε ήδη ε, ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ε, ε, με την Χιλή για τη συμφωνία αυτή ενώ δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει οι γενικότερες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Γενικού Εμπορίου που δεν πρόκειται να ξεκινήσουν παρά μόνο μετά το καλοκαίρι. Και πρόκειται για μια φυσιολογική συμφωνία. Δεν περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει καθόλου εμπορικέ παραχωρήσει. Απλώ περιλαμβάνει την αναγνώριση τη ισοδυναμία των κανόνων παραγωγή και συστημάτων ελέγχου. Και από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε αυτή την ισοδυναμία, ε, τα προϊόντα της χιλής έρχονται χωρίς επιπλέον απαιτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο με του ίδιους όρους και τα δικά μας προϊόντα εξάγονται προς τη χιλή. Το κείμενο της συμφωνίας προβρέπει προβλέπει και ένα μηχανισμό προσαρμογής σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού για τη βιολογική γεωργία έρθουν σε αίσιο πέρας, όπως και ευελπιστούμε. Γιατί θα ήταν δύσκολο να αναθεωρούμε κάθε συμφωνία και μάλιστα χωρίς ε, εγγύηση αποτελέσματος. Οπότε θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη συμφωνία που έχουμε αμοιβαία αναγνώρισης με χώρα της Λατινική Αμερική, αναγνώριση της ισοδυναμίας των βιολογικών προϊόντων, δυνάμει των εντολών που μας έδωσε το 2014 το Συμβούλιο. Γιατί έχουμε σχετική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στόχο μας ήταν να μην περιοριστούμε στη μονομερή αναγνώριση τη ισοδυναμία όπω γινόταν μέχρι τώρα. Όταν μια τρίτη χώρα ζητούσε την αναγνώριση της ισοδυναμίας των κανόνων, εμείς εξετάζαμε το αίτημα και μετά από αναλύσεις και ελέγχους χορηγούσαμε ή όχι την ισοδυναμία. Δεν προ... προβλέπαμε μέχρι στιγμής την αμοιβαιότητα που σε τελική ανάλυση μας ευνοεί. Ευνοεί το δικό μας ε, κλάδο βιολογικής παραγωγής που αυξάνεται ε, με μεγάλους ρυθμούς, γιατί πρόκειται για ένα δυναμικό τομέα τα περισσότερα προϊόντα κατευθύνονται, προορίζονται στην εσωτερική αγορά, αλλά και άλλα προϊόντα θα εξαχθούν, γιατί και οι τρίτες χώρες απαιτούν ποιοτικά βιολογικά προϊόντα, όπως είναι τα ευρωπαϊκά. Και με τέτοιου είδους συμφωνίες θα δώσουμε κίνητρα για την ανάπτυξη του εμπορίου βιολογικών προϊόντων. Τώρα, μιλήσατε για τον αντίκτυπο της συμφωνίας αυτής ε, στη δική μας παραγωγή. Έχουμε πολλά στοιχεία και δεδομένα που αναλύουμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις εξαγωγές της χιλής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ε, το καθεστώς τους, τις ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές και ούτω καθεξής. Είναι στη διάθεσή σας αυτά τα στοιχεία. Αν θέλετε πιο διεξοδικά να τα αναλύσετε, υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα στην Χιλή έχουμε 669 παραγωγούς βιολογικών προϊόντων το 2015 και 65.000 εκτάρια με βιολογική παραγωγή. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 είχαμε 13 εκατομμύρια εκτάρια, ε, σήμερα πολύ περισσότερα, και πάνω από 350.000 παραγωγούς βιολογικής γεωργίας. Οπότε υπάρχει μια σύμμετρη κάλυψη υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συμφωνία αυτή, λόγω της μεγάλης διαφοράς ε, ε, του αριθμού των γεωργών και των γεωργικών εκτάσεων. Επίσης, ε, τέτοιου είδους συμφωνία ανοίγει το δρόμο για άλλες παρόμοιες συμφωνίες που θα παρέχουν αντίστοιχα ωφέλη στους Ευρωπαίους γεωργούς. Αναφέρθηκε πολύ στη συζήτηση το θέμα της ντόπια της τοπικής παραγωγής. Σίγουρα η τοπική παραγωγή είναι πολύ υποφελής ε, και λόγω εγκύτας με τον καταναλωτή και λόγω περιβαλλοντικής προστασίας. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Η βιολογική γεωργία πληρεί συγκεκριμένους κανόνες και ναι μεν πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο ή το μόνο κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη υπάρχουν ε, ουσίες που γίνονται δεκτές ή μερικώς δεκτές. Ε, ισχύουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ε, και προϋποθέσεις για την βιολογική γεωργία που δεν ισχύουν για την συμβατική γεωργία. Και επίσης είναι και το θέμα της επισήμασης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα και σίγουρα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα σημεία. Αν έμεινε κάποια κρεμότητα, πολύ ευχαρίστω να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αποσαφηνίστηκε η κατάσταση, γιατί όντως ε, δίνονται μεγαλύτερα ωφέλη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις δυνατότητες εξαγωγής. Δεν συμβαίνει αυτό συχνά. Και ναι, μεν υπάρχει και το περιβαλλοντικό μειονέκτημα, αλλά οικονομικά υπάρχουν ωφέλη. Σίγουρα από άψη και μεταφοράς ε, η προσπάθεια είναι μεγαλύτερη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη. Ευχαριστώ και η κυρία Γκιλέρα τώρα για να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να ε, πω στη φίλη μου τη Μαρία από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ότι όταν εγώ μιλώ για τη διαδικασία. Δεν εννοούσα ότι ο Επίτροπος Γεωργίας, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, δεν έδειξαν σεβασμό προς, την, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ότι δεν ακολούθησαν τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι προβληματική. Εσείς την ακολουθήσατε. Είναι πολύ καθυστερημένη στιγμή που ζητάτε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εσείς σίγουρα τηρήσατε κατά γράμμα τη διαδικασία. Και ό,τι πληροφορία σας ζήτησα, την έλαβα. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ε, παράλογο και αφύσικο ε, να δίνουμε τόσο καθυστερημένα τη γνώμη μας. Γιατί πολλοί, πολλά λέγονται για τις εμπορικές αλλαγές και η μεγαλύτερη επίκριση που ακούγεται είναι η αδιαφάνεια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα βοηθούσε πολύ πριν την υπογραφή ε, της συμφωνίας της διμερούς ή της πολυμερούς να έχετε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άμα ζητάτε τη γνώμη σας, αφού έχετε ολοκληρώσει τη συμφωνία για να πούμε ένα ναι ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι σωστός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, συμφωνώ. Ακολουθήθηκε η οχι δεν νομιζω οτι ειναι σωστος ο ρόλο του διαδικασία. Ω προ αυτό ήταν άψογη η συμπεριφορά σα. Αλλά η διαδικασία είναι προβληματική. Και έλαβα ό,τι πληροφορία ζήτησα από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Θα ήθελα να το αποσαφηνίσω ότι και ζητώ συγγνώμη αν αυτή ήταν η εντύπωση που δημιούργησε η Μαρία Άγχελες. Εγώ δεν αφισβήτησα ότι τηρήσατε πιστά τη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι η διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που οφείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε συμφωνίες δηλαδή εμπορικές. Και μια και έμεινε λίγος χρόνο να ολοκληρώσω τα βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές. Υπάρχει το θέμα της εγκύτητας, υπάρχει η ανάγκη πρόθεση της τοπικής παραγωγής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα και στόχοι και χρήσιμα μέτρα για να έχουμε ντόπια προϊόντα κοντά στον καταναλωτή, φρέσκα προϊόντα εποχιακά και να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά δεν θα πρέπει να το μπερδεύουμε αυτό με το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ νομοθετούμε με την συμφωνία αυτή και ρυθμίζουμε τις εμπορικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες για τα βιολογικά προϊόντα. Και εγώ προτιμώ να έχουμε κανονιστική διαδικασία για τα βιολογικά προϊόντα σε μια εμπορική συμφωνία παρά να μην έχουμε καθόλου τέτοια ρύθμιση και συμφωνία. Γιατί ε, εμπορικές σχέσεις θα υπάρχουν, είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι. Γι' αυτό και εγώ προτιμώ να έχουμε ρυθμισμένη διαδικασία, κανονιστική, σε μια συμφωνία που να διέπει και τα βιολογικά προϊόντα, παρά να αφήσουμε το ζήτημα αριθμιστό. Και υπάρχει μία πρόοδος, γιατί οι δικές μας αυστηρότερες προδιαγραφές και οι δικοί μας αυστηρότεροι κανόνες αναγνωρίζονται ε, για τα βιολογικά προϊόντα σε συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Και αυτή είναι και η καινοτομία. Βέβαια, ίσως υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για την πραγματική ισοδυναμία, αλλά προτιμώ στις εμπορικές μας σχέσεις να ισχύουν κανόνες από το να είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτά ευχαριστώ και για όσοι ενδιαφέρονται, αύριο στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα συζητηθεί έκθεση της για τη συμφωνία αυτή. Μάλιστα. Α, έτσι έχει η διαδικασία. Εμείς πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Η συγκέντρια προτείνει ναι για τη συμφωνία. Νομίζω ότι από τη συζήτηση έγινε αντιληπτή η κατάσταση σε, αυτή την, ε, σε αυτό το μικρό μερίο της αγοράς που καλύπτει η βιολογική γεωργία. Ευχαριστώ το, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Μέχρι τις 5 Μαΐου, στη μία η ώρα μπορούν οι συνάδελφοι να καταθέσουν τροπολογίες όπως προβλέπει η διαδικασία. Περάμε τώρα στο επόμενο θέμα, την παρουσίαση της ε, έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας παρουσιάσει ο Διευθυντής ε, Μιχαήλ Ντουμήτρου από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για την εφαρμογή των υποχρεώσεων ε, των περιοχών οικολογικής εστίασης στο καθεστώς πράσινων άμεσων πληρωμών. Στόχος ήταν να βελτιώσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων στη Γεωργία μέσω της, μέσω της των πληρωμής άμεσων ενισχύσεων που έχουν σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, πέραν της ψησποράς και της διατήρησης μόνιμων βοσκοτόπων η οικολογικοποίηση απαιτεί από τους γεωργούς να κρατήσουν 5% των αρρώσιμων ε, γεωργικών εκτάσεών τους για περιοχές οικολογικής εστίασης. Και μάλιστα αυτή η πρόοδος εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο πληρούνται με τις ε, μεταρρυθμίσεις του 2013 ή υποχρεώσεις για την οικολογικοποίηση και τη θέσπιση περιοχών οικολογικής εστίασης. Θα ακούσουμε τα πορίσματα της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο ε, εκπληρώθηκαν αυτές οι υποχρεώσεις του 5% των γεωρικών εκτάσεων για τις ε, περιοχές οικολογικής εστίασης και το κατά πόσο αξιοποιήθηκαν τα σχετικά κονδύλια. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τη γενική Διεύθυνσης Άγκρη, ο κύριος Μιχάηλ Ντουμίτρου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε κυριε. και κύριοι, όπω ανέφερε και ο Πρόεδρος, η Επιτροπή στη συλλογική της σύνθεση στις 29 Μαρτίου υιοθέτησε τη γνωμοδότηση για την υιοθέτηση των περιοχών οικολογικής εστίασης που είναι ένας ε, νέος παράγων ε, οικολογικοποίησης. Πρόκειται για μια νομική υποχρέωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία η οποία δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται. Μήπως να έρθετε στο Προεδρείο, ίσως είναι καλύτερο. Όχι, όχι, θα με βοηθήσει κάποιο για να προχωρήσουν οι διαφάνειες, αλλά συνεχίσω όσο η συνάδελφος ασχολείται με, το, με τα εποπτικά μέσα. Λοιπόν, πρόκειται και μια υποχρέωση που προκύπτει από τον βασικό κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι το Μάρτιο του 2017, λοιπόν, έπρεπε να καταθέσουμε μια έκθεση για τις περιοχές οικολογικής εστίασης και ταυτόχρονα μια πρόταση για ενίσχυση των ποσοστών τους από 5 σε 7%. Η Επιτροπή είχε εντωμεταξύ αποστείλει την πρόταση στη γραμματεία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έτσι φαντάζομαι ότι θα έχετε στα χέρια σας την πλήρη έκθεση. Εν εδώ παρουσιάζουμε μια επισκόπηση και αξιολόγηση των πρώτων ε, δύο ετών της υλοποίηση αυτής της προπόθεση και μια προκατακτική αξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών συνεπειών. Στόχος λοιπόν της σημερινής μου παρουσίας ήταν να σα εκθέσω τα κύρια αποτελέσματα αυτής τη πρώτη διετία εφαρμογή των περιοχών οικολογική εστιαση ΠΟΕ, και όπω είπα αποτελεί συνέχεια της ανάλυση που κάναμε πέρσι στο πλαίσιο τη οικολογικοποίηση ύστερα από ένα έτος εφαρμογής που έχουμε υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σα δώσω προκατακτικές ε, εικόνες από τις πιθανές ε, ε, συνέπειε για το περιβάλλον των ΠΟΕ και τις αύξησή του. και τις και την πρόταση συγκεκριμένα για αύξηση από 5 σε 7% των ΠΟΕ. Είναι αναλυτικό έργο, συλλέγει τα δεδομένα, η έκθεση από την περσινή ε, επισκόπηση, η οποία, υπενθυμίζω, εστιάστηκε στο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, το δυναμικό παραγωγής, και την πρόταση του Απριλίου 2014 για τη ΣΠΟΕ. Ο Φιλ Χόγκαν, ε, Επίτροπος, άλλωστε περιέλαβε τις προτάσεις αυτές στις, ε, στη δέσμη για απλούστευση που προτάθηκε σε σχέση με την οικολογικοποίηση, με μεγάλη έμφαση στις ΠΟΕ, σε τροποποίηση της κατεξουδότησης πράξης 639 του 2014 υιοθετήθηκε πριν τις 14 Απριλίου, ε, Φεβρουαρίου του 2017 και όπως είπα έχει περάσει από το συλλογικό, την Επιτροπή στη Συλλογική της Σύνθεση. Στόχος λοιπόν ΠΟΕ. Στόχος τους είναι να διαφυλάξουν και να βελτιώσουν τη βιοπικιλότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπως είχε ζητηθεί να υπάρχει αυτός ο περιβαλλοντικός δεσμός της διαφύλαξης της βιοπικιλότητας αλλά και της προστασίας των εδαφών, των υδάτων και του κλίματος. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει αυτή η διάταξη η οποία λέει ότι οι εκμεταλλεύσεις που έχουν πάνω από 15 εκτάρια έκταση πρέπει το 5% να ε, ε, παρουσιάζεται ως περιοχή οικολογικής εστίασης με διάφορες, με μια μεγάλη ποικιλία επιλογών. Ε, μπορεί να είναι είτε περιοχές σε αγρανάπαυση, είτε ζώνες ανάσχεσης, είτε ε, βελτίωση των εδαφών, ε, καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο, και Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ελευθερία για τα κράτη να ορίσουν αυτή την ε, γκάμα των επιλογών με βάση τις βέλτιστες ε, δυνατότητες και βέβαια για τον Γεωργό αντίστοιχα, ο οποίος θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ΠΟΕ ΕΕ από την, με βάση τον εθνικό κατάλογο. Υπάρχει ένας παράγων αναμονής, πρέπει να επισημάνω, ο οποίος έχει να κάνει με τον ε, βαθμό συμβολή στη βιοποικιλότητα της κάθε ΠΟΕ και τα οικολογικά ωφέλη. 0,3 για τις, ε, για τις επίσπορες καλλιέργειες και για τις ε, καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο. Ε, για να κοιτάξουμε λίγο τα στοιχεία, ύστερα από δύο χρόνια υλοποίησης του συστήματος, βλέπετε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλα τα κράτη 2015 και για τα περισσότερα, για το 2016-2019 κράτη συγκεκριμένα βλέπετε μικρή διακύμανση μεταξύ των δύο ετών, είτε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σύστημα, είτε τα κράτη-μέλη, στον τρόπο με τον οποίο οι γεωργοί ε, πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Ε, το 70% μεγάλη πλειονότητα της αρρώσιμης γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγεται στην υποχρέωση ΠΟΕ. Υπάρχει η εξαίρεση, όπως είπα, ε, που έχει να κάνει με το υπόλοιπο ποσοστό και είναι οι βιολογικές καλλιέργειες, μικρές καλλιέργειες κάτω από 15 εκτάρια κτλ. 8 εκατομμύρια λοιπόν εκτάρια στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 13% ε, των εκτάσεων που είχαν υποχρέωση ΠΟΕ είχαν χαρακτηριστεί ΠΟΕ, άρα έχουμε με βάση τη στάθμιση ένα 10% των εκτάσεων. και να καταλήξω λοιπόν έχουμε το διπλάσιο από το 5% που απαιτούσε η νομοθεσία με βάση τη νομοθεσία με βάση την έκταση της ε, εκμετάλλευσης και δεν αλλάζουν οι τάσεις αυτές, παραμένουν σχετικά σταθερές. Ας δούμε τώρα τι είδου οικολογικές ε, περιοχές οικολογικής εστίασης έχουν επιλεγεί από τις ε, παραγωγικές περιοχές, 92,5% του συνολικού, των συνολικών ΠΟΕ, βλέπουμε είτε καλλιέργειες που δεσμεύουν άζωτο με το μεγαλύτερο ποσό 39%, είτε αγρανάπαυση με 38,5%, είτε επίφορες, επίσπορες καλλιέργειες 15%, δασικές καλλιέργειες ή γη με χαρακτηριστικά τοπίου ή ζώνες ανάσχεσης με ένα συνολικό 4,5%. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ε, αναπτύσσεται αυτή η κατανομή των ειδών ΠΟΕ ανακράτος Έχουμε διαφορετική εικόνα, ανακράτος μέλος. Ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη, όπως βλέπετε, έχουν ξεπεράσει το 5% σε ΠΟΕ. Πολλά φτάνουν και πάνω από το 10% και επιπλέον η σύνθεση των ΠΟΕ ανακράτος μέλος έχει διαφορετική απεικόνηση πάλι, ανάλογα και με αυτά τα οποία σας ε, είπαμε την προηγούμενη διαφάνεια, η αγρανάπαυση, οι επίσπορες και οι καλλιέργειες που δεσμεύουν ε, άζωτο, που εμφανίζονται σαν ένα, επιπλέον του 5%, το πετουμένο 5% ποσοστό ή μπορεί να συμβάλλουν κατελάχιστον στην κάλυψη της απέτησης για 5%. Άλλοι τύποι των ΠΟΕ όπως υγεία, χρανάπαυση θα αρκούσαν για την κάλυψη του ποστού 5% στα προστορα μελη Ωστόσο το ποσοστό των καλλιεργειών δέσμευσης αζότου είναι πιο χαρακτηριστικό, ε, πιο σημαντικό σε αυτές τις χώρες που ξεπερνούν το 5% σε ΠΟΕ. Και περαιτέρω. Τι καινούριο μας φέρνει αυτή η έκθεση σχέση με προηγούμενες. Και αυτό είναι η αξιολόγηση των πιθανών ωφελών ε, των ΠΟΕ και σε βιοπικιλότητα αλλά και σε υπηρεσίες στα οικοσυστήματα. Σε σχέση λοιπόν με την προηγούμενη επισκόπηση πάμε περαιτέρω και εξετάζουμε πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες ανάλογα με τον τρόπο που υλοποιήθηκαν οι ΠΟΕ μέχρι τώρα. Σημειώνω ότι πρόκειται για μια θεωρητική ε, αξιολόγηση με βάση τη σχετική φιλολογία αλλά και πρότυπα του Κοινού Κέντρου Ερευνών υπολογισμό ΠΟΕ, ε, ε σύστημα υπολογισμού ΠΟΕ όπως το λέμε που μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη την σύνθεση σε περιφερειακό επίπεδο και τις επιλογές που για όλους τους γεωργούς μιας περιφέρειας σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3 οι προσωμιώσεις μας μας δείχνουν ότι ανάλογα με την ΠΟΕ αλλάζουν και οι επιλογές και οι αναλύσεις δείχνουν ότι όλες οι ΠΟΕ όλοι οι τύποι ΠΟΕ και η σύνθεσή του σε επίπεδο υποπεριφερειακών ΑΤΣ3 μπορούν να φέρουν θετικό αντίκτυπο στη βιοπικιλότητα. Διαφορετικού όμως επίπεδου αντίκτυπο. Με μεγαλύτερο δυναμικό σε θετικό αντίκτυπο για την σύνθεση με χαρακτηριστικά τοπίου σε μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 50% του συνολικού της ΠΟΕ και δεύτερο επίπεδο, αγρανάπαυση με ποσοστό πάνω από 70%. Χαμηλότερες επιδόσεις είχαν ε, οι εμβόλυμες, οι εμβόλυμες ε, καλλιέργειες. Αλλά δεν έχουμε μόνο το, την επιλογή που ε, έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν ότι η βιοπικιλότητα, η υπηρεσία στα οικοσυστήματα έχουν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης ανάλογα με τον τύπο ΠΟΕ. Ε, παραδείγματι, η κάλυψη εδαφών για αγρανάπαυση, τα διαφορετικά ε, είδη καλλιεργειών για τις επίσπορες ή εμβόλυμες καλλιέργειες ή για τις καλλιέργειες που έχουν κρατές δεσμεύσεις αζότου ή περίοδοι που ε, χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι, τα χημικά που χρησιμοποιούνται, η δε περίπτωση και οι ζώνες ανάσχεσης αλλά και ε, όταν έχουμε ε, περιοχή αγρανάπαυσης με μεγάλα ποστά σε λουλούδια παραδείγματι μπορεί αυτό να έχει πολύ, καλές, ε, πολύ θετικό αντίκτυπο σε σχέση με την επικονίσιαση όταν δεν χρησιμοποιούνται ζυζανιοκτώνα σε περιοχές αγρανάπαυσης έχουμε θετικό αντίκτυπο ιδιαίτερα όταν συμπίπτει αυτό με την περίοδο ε, ζευγαρώματος ε, των ε, πτηνών. Τώρα, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, και εδώ είναι το κύριο συμπέρασμα της επισκοπησής μας. Προτείναμε αλλαγές πρόσφατες στην οικολογικοποίηση Ω ένα σημαντικό βήμα για καλύτερες διαχειριστικέ πρακτικές και απλούστευση βέβαια των μέτρων. Και αναφέρομαι σε μια περίοδο εναλλαγής μεταξύ της, ε, των εμβόλυμων καλλιεργιών και των, ε, και των εκτάσεων σε αχρανάπαυση και επίσης ε, θέλω να σταθώ λίγο στην πρόταση για αύξηση από 5 σε 7%. Δεν βλέπουμε λόγο να αυξηθούν οι ΠΟΕ για τους λόγους που σας εξέτασα νωρίτερα, από το 5% στο 7%, αλλά εάν υπήρχαν εναλλαγές στις επιλογές του τύπου ΠΟΕ, των γεωργών και τις πρακτικές διαχείρισης, θα είχαμε πολύ καλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν ως προς τις εκτάσεις είμαστε ικανοποιημένοι ε, και ως προς τις επιλογές θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα της διαχείρισής τους. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, σε αυτή τη συζήτηση να ακούσουμε τους συνέδρους. Πρώτα ο κύριος Ντες. Φανταζόμουν θα το ζητήσει σε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για αυτήν την παρουσίαση η οποία απέχει νομίζω πάρα πολύ από το τι γίνεται στην πράξη. Ελπίζω να μην ακούγε κανένα αγρότης, πάλι θα απογοητευτεί από την Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να αξιολογείτε τις πρακτικές ε, θετικές και αρνητικές. Κοιτάξτε, εγώ διαπιστώνω ακριβώς στη δικιά μας την περιφέρεια πως αυτές ακριβώς οι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάτε για το ξαναπρασίνισμα και όταν μιλάτε ακριβώς για τις ζώνες ε, οι οποίες είναι κοντά στα δάση και δεν ε, καλλιεργούνται. Πράγματι είναι ιδιαίτερος οικολογικές, αλλά είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση ώστε δεν ασχολούνται καθόλου οι αγρότες από το να κάνουν ένα λάθος στην ε, εφαρμογή. Εν τω μεταξύ μιλάτε για τα φυτά εκείνα τα οποία δεσμεύουν το άσδομα είναι 93% των φυτών ε, δεσμεύουν το άσδο. Εν τω μεταξύ, τι καταλήγουμε, καταλήγουμε στο να εισάγουμε ψόγια από την ε, Νότια Αμερική και έχουμε άλλο ένα εκατομμύριο τόνου. Ελπίζω λοιπόν να διορθωθούν αυτά τα λάθη και να συνεχίσουμε να μπορούμε στο μέλλον να καλλιεργούμε πρωτεϊνούχα φυτά στις ε, περιοχές αυτές γιατί είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα πρωτεϊνούχα φυτά και δεν πρέπει ε, να ξεχνάμε ότι δεν έχουν την ίδια ανθοφορία με τα, άδεια, με τα άλλα φυτά. Πρέπει λοιπόν να συζητείτε το θέμα επαρκώς και με κάποια νομίζω ικανότητα και σχέση με την πραγματικότητα γιατί πραγματικά σπάνια έχω δει παρουσιάσεις που να είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Συμφωνήσαμε 1,5 λεπτό καθένας, ο κύριος Λουαζό. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εγώ όπως και περισσότεροι Γεωργοί, με τη στήριξη των συνδικάτων, των συνεταιρισμών τους, είμαστε κατά της κατεξοδότηση πράξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει να επιβάλλει για το 2018 επιπλέον περιορισμούς για την οικολογικοποίηση, σαν να μην είχαμε αρκετούς περιορισμούς ήδη. Και μάλιστα το μέτρο που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους γεωργούς είναι αυτό που ζητά απαγόρευση οποιαδήποτε εφαρμογή φυτογειονομικού προϊόντος σε καλλιέργειες ψυχανθών, ε, κυρίως αυτό που εξομοιώνονται με περιοχές οικολογικής εστίασης. Η υποχρέωση αυτή θα μειώσει de facto της ε, γεωργίας εκτάσεις καλλιέργειας ψυχανθών και επίσης ε, θα αυξήσει την αύξηση των γεών υπογρανάπαυση. Ελπίζω να έχετε επίγνωση αυτού του γεγονότος γιατί θα αναγκαστούμε έτσι να εισάγουμε τις πρωτεϊνούχες, ε, τα πρωτεϊνούχα προϊόντα που μας λείπουν. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ο κύριος Κάρθη για 1,5 λεπτό. Thank you, Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί έχασα την παρουσίαση, αλλά την έχω διαβάσει. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε αυτή τη στιγμή ότι οι απαιτήσει πρασινίσματο, όπω λέγεται τη Κομισιόν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε πολλέ χώρες ε, δεν προβλέπουν ευελιξία και την ποικιλομορφία που υπάρχει σε διάφορε χώρες και βλέπουμε ότι η Κομισιόν ε, θα πρέπει να δώσει αυτή την ευελιξία γιατί εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έχουν αντίκτυπο τα μέτρα. Παραδείγματο χάρη στην Ιρλανδία, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ε, κάποια μέτρα ισοδυναμία για να λάβουμε υπόψη ε, τα λίγα είδη τα οποία μπορούν να καλλιεργούν οι γεωργοί. Τώρα υπάρχουν προσπάθειες ε, για να υιοθετήσουν το πρόγραμμα. Η Γεωργία, αλλά μόλι 25 γεωργοί συμμετείχαν στο πρόγραμμα ισοδυναμία πέρσι. Ε, Νομίζω είναι σαφές το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και το μιλάμε για τα EFA. Οι δηλώσεις ε, αυτές ε, ήταν πραγματικά τέρατα γραφειοκρατίας ε, και διοικητικού βάρους και βεβαίως σημαίνει ότι υπήρχαν και βαριά πρόστιμα. Θα πρέπει επίσης να είναι πιο αναλογικά, αναλογικά με πρόστιμα και να απλοποιηθούν οι σχετικές ε, δηλώσεις ε, των γεωργών. Έτσι θα μεταρρυθμίσουμε αρκετά το σύστημα, κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Η αντίδραση των περισσότερων εδώ στην παρουσίαση είναι η λέξη περιπλοκή. Είναι πολύ περιπλοκό το σύστημα και νομίζω πως το βασικό λάθος ήταν ότι προσπαθήσαμε να το βάλουμε στον πυλώνα 1. Φοβάμαι ότι ο πυλώνας 1 θα έπρεπε να έχει μείνει μόνο για την χρηματική στήριξη των γεωργών. Και μετά να έχουμε ένα δεύτερο πυλώνα, όπου θα έχουμε όλα αυτά τα διάφορα συστήματα και το κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει τι θέλει. Μετά, από εκεί συνεχίζουμε και μιλάμε για αγρανάπαυση. Τις παλιές καλές μέρες θα λέγαμε, όταν δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε τα ζυζάνια, η αγρανάπαυση ήταν ακριβώς μέρος ότι αλλάζαμε τις καλλιέργειε και για να, είναι, για να υπάρχει αγρανάπαυση έπρεπε να οργώσουμε τέσσερις φορές το χρόνο. Βεβαίως το όργωμα σημαίνει ενέργεια και ανακατεύει και το χώμα και δεν είναι τόσο καλό για το περιβάλλον θα λέγει κανείς, αλλά αναρωτιέμαι αν περισσότερος κόσμος γνωρίζει το τι σημαίνει αγρανάπαυση. Οπότε τι κάνουμε απλά αφήνουμε το χωράφι ε, ως έχει από την τελευταία σοδιά. Τελικά θα έρθουν μόνιμα ζυζάνια, δηλαδή όπως το χωρεί αυτή η γη από καλλιεργήσιμη και τελικά υπάρχει και μία αντίφαση εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πρωτεϊνούχα φυτά. Εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τις εισαγωγές. Οπότε θα μπορούσαμε να, να, να πούμε εντάξει, αν θέλετε κάποιο υποκατάστατο πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Ε, το οποίο είπαν, αλλά μετά είπαν Α, όχι, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υλικά φυτοπροστασίας, πρέπει ουσιαστικά να είναι βιολογική καλλιέργεια χωρίς παραπάνω όφελος, οπότε θα χάσουν λεφτά. Βεβαίως μπορούν, μπορούν ε, να καλλιεργούν ε, μόνο κατά 50% οι γεωργοί ε, και βεβαίως ε, τι θα σημαίνει αυτό, τελικά θα χάσουν. Εάν θέλουμε πρώτα οι νούχες σοδιές στην Ευρώπη, πρέπει να τις στηρίξουμε. Σωστά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι νέες τεχνολογίες όμως αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά αυτή τη συχνή άρρωση. Η κυρία Μίλλερ. Ναι κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για το ότι ο κύριος Ντες ήρθε τώρα στους ε, φιλελεύθερους και νομίζω θα νιώσει αν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις δηλώσεις της. Ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα όσον αφορά το γιατί ε, βρεθήκαμε με αυτήν την πρόταση. Διαπιστώνουν μόνοι τους ότι δεν είναι αναγκαία μία αύξηση από το 5% στο 7% αλλά θέλουν να βελτιωθεί η ποιότητα των ε, εκτάσεων οικολογικής ε, προτεραιότητας. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι εκτάσεις να μην ε, θεωρηθούν βιολογικές εκτάσεις, αλλά απλές αρωτρές εκτάσεις, τις οποίες σε συνεργασία με τους γεωργούς θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε την βιοπικιλότητα. Νομίζω ότι καταφέραμε αυτό να γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και θα πρέπει ακριβώς ε, να έχουμε κατανοώ αυτό το οποίο έγινε για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε μόνοι μας πρωτεϊνούχα φυτά και θα πρέπει μία φορά την άνοιξη να χρησιμοποιούνται ζυζανιοκτώνα. Και μετά τέλος, και όταν έρχονται μετά οι μελισσοκόμοι και λένε ότι χαίρονται ακριβώς για την καλλιέργεια ψυχανθών και αναγνωρίζουμε ότι δεσμεύουν και άζωτο, τότε για μένα νομίζω τελειώνει. Εδώ πέρα το ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει, να δούμε ποια είναι η προσθέμενη αξία. Πρέπει να υπάρξει μια απλούστευση του λεγόμενου πρασινίσματος. Δηλαδή, κατά πόσο συνεισφέρει η απαγόρευση των ζανιοκτώνων στην απλοποίηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ντελέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω ένα σχόλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευτυχώς ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έχει νόημα να περάσουμε στο 7%, θα παραμείνουμε στο 5%. Είναι ήδη αρκετό το 5%. Να αφήσουμε του γεωργού να ασκούν τη γεωργική του δραστηριότητα. Το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμά να το κάνουν, από ότι εμεί ε, οι πολιτικοί ή οι συνεργάτε ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει με πρόσχημα την απλούστευση να πολλαπλασιάζουμε την περιπλοκότητα είπαμε ότι η αγρανάπευση επιτρέπει την ανάπτυξη κάποιων φυτών, όχι όμως μόνο των φυτών, αλλά και των ζυζανίων. Και όταν υπάρχουν ζυζάνια θα πρέπει να μπορεί ο Γιώργος να τα ξεχερσώνει. Ε, αλλιώς δεν θα μπορέσει να περάσει την επόμενη καλλιέργεια, αν δεν έχει ε, ξεριζώσει τα ζυζάνια. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει αυτές, αυτή η αγρανάπαυση τουλάχιστον να προσελκύει τις ε, μέλισσες με τα φυτά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ε, τη γύρη που χρειάζονται και ακριβώς η έλλειψη γύρης οδηγεί μερικές φορές στη μεγαλύτερη θνησιμότητα των μελισσών. Ευχαριστώ κύριε Κέστιγκερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για το ότι απέδειξε ότι τα πράγματα δεν γίνονται απλώς τώρα, αλλά ε, όλο και πιο περίπλοκα για τους γεωργούς, ειδικά στην εφαρμογή. Εγώ από μια χώρα η οποία ε, εδώ και δεκαετίες ε, έχει στραφεί στην καλλιέργεια χωρίς γενετικά τροπημένους οργανισμούς και παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω τι θέλει αυτή η πρόταση της Κομισιόν. Ήμουν και διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τελευταία μεταρρύθμιση και υπήρχε κάποιος λόγος για τον οποίο μιλούσαμε για ζώνες οικολογικής προτεραιότητας και όχι βιολογικής καλλιέργειας. Είναι δεδομένο πράγματι ότι συμφωνήσαμε σε αυτά τα φυτά τα οποία δεσμεύουν άζωτο για να προωθήσουμε αφενός και την οικολογία αλλά να υπάρχει και ένα κίνητρο για τις εκμεταλλεύσεις. Αυτό το ξεχνούν πάρα πολύ οι ειδικοί και θα ήθελα να πω ότι είμαστε, θα περίμενα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να είναι στο πλευρό των αγροτών γιατί βεβαίως η απαγόρευση αυτή σημαίνει και απώλεια εισοδήματος. Το είδαμε αυτό νομίζω και στα νούμερα. Υπάρχει μία υιοθέτηση, λειτουργεί και δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει αλλαγή μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και θα ήθελα να παρακαλέσω από την Κομισιόν να το ξανασκεφτεί. Ο κύριος Δάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρουσίαση της έκθεσης ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολλό δε μάλλον που η Γαλλία δεν περιλαμβάνει τις χώρες που αναλύθηκαν, γιατί η κυβέρνηση δυστυχώς δεν εφάρμοσε σωστά την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πέραν όμως αυτών των εθνικών ε, στοιχείων, ε, διαπιστώνω ότι μια καλή ιδέα μπορεί να γίνει μια τρύπα μέσα στο νερό. Γιατί σε ό,τι αφορά την οικολογικοποίηση, που είπαμε πριν από πέντε χρόνια ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα ιδέα και ανταποκρίνεται σε ένα κοινωνικό αίτημα, ε, είχαμε συμφωνήσει να συμπαρασταθούμε σε μια θετική προσέγγιση των γεωργών. Και αντί να κάνουμε κάτι τέτοιο, θεσπίσαμε και πάλι μια πολιτική περιορισμών και ελέγχου. Οπότε δεν θα πρέπει να εκπλησώμεθα που οι γεωργοί όλο και περισσότερο αρχίζουν και γίνονται επιφυλακτικοί απέναντι στις πολιτικές μας και εχθρικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε πολιτικές θετικής συμπαράστασης ε, των γεωργών και να ξεφύγουμε αυτή την ε, υπερβολική περιοριστική πολιτική που μας ε, οδηγούν προς μια προαναγγελθής καταστροφή. Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την έκθεσή της. Με ενδιαφέρουν τα δυνητικά ωφέλη. Είστε σίγουροι για αυτή την αξιολόγηση που κάνατε τη οικολογικοποίησης, που είναι μια θεωρητική επιχάρτου. Εγώ θα ήθελα μια ουσιαστική αξιολόγηση της οικολογικοποίησης. Σε ό,τι αφορά τα πορίσματα, είπαμε ε, αν το 5 το 7% είναι ε, χρήσιμο. Δεν χρειάζεται να το γράψουμε στην έκθεση, αλλά έχει φανεί ότι η αύξηση ε, των περιοχών οικολογικής εστίασης προέρχονται κυρίως από τις επίσπορες καλλιέργειες, τη γη υπογρανάπαυση και τις αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά το πρώτο 5% που ήδη υπήρχε και που αφορά κάποιες ζώνες ανάσχεσης ε, ή κάποιε ε, μη καλλιεργήσιμε ζώνε στα περιθώρια των γεωρικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, ε, κάτι που ενδιαφέρει τους ε, συναδέλφους για τη χρήση φυτοφαρμάκων στις αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες. θα ήθελα να το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πώς θα α, αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στο μέλλον, γιατί για κάποιο λόγο μπήκε αυτό το σημείο στη σημερινή φάση της οικολογικοποίησης. Στο μέλλον όμως τι μορφή θα πάρει. Ευχαριστώ κύριος Δεκάστρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και σύντομα γιατί πολλά τα κάλυψαν ήδη οι συνάδελφοι. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη και να υπενθυμίσω τη σημασία του να μην διακοπεί αυτή η καλή πρακτική που έχουν οι γεωργοί μας, δηλαδή μέρος της γεωργικής τους ε, ε, έκτασης να το καλύπτουν με ψυχανθή πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο. Με τα, φυτοφάρμακα θα χάναμε δεκάδες χιλιάδων εκταρίων στη χώρα μου ιδιαίτερος μπορούμε να έχουμε καλλιέργειες εκατοντάδων χιλιάδων νεκταρίων χωρίς ε, ε, γενετικά τροπημένους οργανισμούς, πρωτεϊνούχων ε, ψυχανθών και θα ήθελα ή μη τι άλλο να εξασφαλιστεί μια παρέκκληση, μια εξαίρεση για εκείνες τις καλλιέργειες οι οποίες βελτιώνουν το έδαφος. Ευχαριστώ και πολύ κυρία Αγγελέρα. Και εγώ συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των προλυσάντων. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα στις περιοχές οικολογικής ε, ε, εστίασης να απαγορευτούν τα φυτοφάρμακα. Δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο, ούτε το βήμα που θέλετε να κάνετε με την πρόταση αλλαγές. Γιατί πρόκειται για ζώνες, αρρώσιμες εκτάσεις, που, στις οποίες θέλουμε βελτίωση της βιοπικιλότητας. Και αυτό γίνεται, είναι ορατό. Και όπως είπε ο κύριος Δεκάστρο, είναι πολύ θετικό το έργο των γεωργών στις περιοχές οικολογικής εστίασης και των γεωργών και των κρατών μελών. Γιατί να αλλάξουμε τώρα ε, την κατάσταση και να απαγορεύσουμε τα φυτοφάρμακα στις περιοχές οικολογικής εστίασης. Αυτό δεν δικαιολογείται με τίποτα. Γιατί οι περιοχές οικολογικής εστίασης απλώς ευνοούν τη βιοπικιλότητα. Δεν ε, ασκούν βιολογική παραγωγή. Γιατί λοιπόν να απαγορεύσουμε τα φυτοφάρμακα. Δεν ξέρω αν ε, η απαγόρευση αυτή είναι μια χειρονομία προς ποιους κύκλους δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν βλέπω να δικαιολογείται μια τέτοια απαγόρευση. Γιατί αναγνωρίζεται το θετικό έργο. μέχρι στιγμής είχαμε επιτρέψει τα φυτοφάρμακα στις ε, περιοχές της οικολογικής εστίασης και τώρα θέλετε να το απαγορεύσετε γιατί, δεν είναι πια της μόδας. Νομίζω ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε το θετικό έργο και την υλοποίηση του στόχου της αύξησης της βιοπικιλότητας δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε τίποτα άλλο και δεν δικαιολογείται η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων. Υπάρχει μεγάλο αίτημα για, φυ... για πρωτεϊνούχα φυτά και θα είναι κρίμα να περιορίσουμε αυτή την παραγωγή. Δεν βλέπω καμία αιτιολόγηση αυτή τη πρόταση. και δεν την καταλαβαίνω καθόλου. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Γενική Διευθυντά, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ πρώτα στην έκθεση, γιατί αυτό ήταν ο ρόλος μου, να παρουσιάσω τα πορίσματα της έκθεσης. αυτό βεβαίως, μια έκθεση τέτοια που είναι κομμάτι μια διαδικασία αναθεώρηση και αξιολόγηση διαφορών στοιχείων τη κοινή γεωργική πολιτική να οδηγεί σε συμπληρωματικά στοιχεία, όπω πρόταση για απλούστευση, που υιοθετήθηκε με την κατεξουδότηση πράξη για την οικολογικοποίηση. Προσπαθούμε λοιπόν να σας προσφέρουμε μια εικόνα, μια, ένα στιγμιότυπο της κατάστασης ύστερα από τον πρώτο και το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του συστήματος, πώς τήρησαν τις προϋποθέσεις πρώτα οι και μετά τα κράτη. Και μιλούμε με δεδομένα, με γεγονότα, με βάση πληροφορίες που μας διέθεσαν τα κράτη-μέλη καταγράφουμε τα στιγμιότυπα αυτά με 90% των επιλογών για τις παραγωγικές ή δυνάμει παραγωγικές περιοχές που έχουν επιλέξει οι γεωργοί. Του τουλεχθέντος το άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με τις εκτάσεις τοπίου που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θέλαμε να δώσουμε και κίνητρα και να ε, αφαιρέσουμε από το σύστημα συστήματα που τώρα παρεμποδίζουν τον ε, γεωργός προς την επιλογή αυτής της ε, λύσης της γης με χαρακτηριστικά οποίο Έτσι λοιπόν όχι μόνο η απαγόρευση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών, ε, έχουμε να κάνουμε μια δέσμη μέτρων με πολύ περισσότερα αυτού στοιχεία. Με ακούτε. Μάλιστα. Και σε σχέση με την απέτηση αξιολόγηση του αντικτύπου. Θεωρητική, προς το παρόν, όπως είπα, η στραπεπισκόπηση και αξιοποίηση της φιλολογίας και δεν, ικανοποιημένη, δεν ικανοποιητική για, την, για το επίπεδο τη δική μα τη επισκόπηση, αλλά όπως είπα και ότι είναι μόνο θεωρητική, άλλα στοιχεία δεν έχουμε. Το σύστημα υπολογισμού, ε, η αριθμομηχανή, θα έπρεπε να δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία και ελπίζουμε ότι στο τέλος του έτους όταν έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη χρονιά επισκόπησης της οικολογικοποίησης και μετά βέβαια πάλι την, τα στοιχεία που μας έχουν δώσει τα κρατη για τις ΠΟΕ θα έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη χρήση και τα εργαλεία αυτού του εργαλείου για την κοινωνική πολιτική. Όπως είπα, κύριος στόχος ήταν η προστασία της βιοποικιλότητας και έτσι η εισαγωγή της απαγόρευσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών σε ε, παραγωγικές ή δυνάμικα παραγωγικές καλλιέργειες είχε σαν στόχο ακριβώς αυτό το στόχο να ενισχύσει. Η ΚΑΠ έχει μεγάλο περιθώριο για προστασία και υποστήριξη μάλλον των ε, ψυχανθών, γιατί έχουμε να κάνουμε 80 εκατομμύρια εκτάρια αρρώσιμης γης με ένα 40% τουλάχιστον. Και εδώ έχουμε την αξιολόγηση των καλλιεργιών που δεσμεύουν άζωτο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο δυναμικό για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην μπερδέψουμε το στόχο της παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης στην Ευρώπη με τον στόχο της προστασίας της βιοποικιλότητας, για τον οποίο έχουμε αναπτύξει εργαλεία και για τα οποία προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς τα αξιοποιούν τα κράτη-μέλη και για τα οποία θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε κέντρα στα κράτη-μέλη για να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα υφιστάμενα εργαλεία, ώστε να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους της ΚΑΠ για την συγκεκριμένη αυτή περίοδο. Βεβαίως. Μπορούμε να δούμε σε ποιο βαθμό η δέσμη μέτρων ε, για την απλούστευση φέρει τα αποτελέσματα ακριβώ αυτά της απλούστευσης. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν απλουστευμένες ε, λύσεις και μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τον γεωργό να χρησιμοποιήσει γη με χαρακτηριστικά οποίο Αν αφήσουμε τις μικρολεπτομέρειες, τη διάσταση του φράχτη ή άλλα στοιχεία της γης με χαρακτηριστικά τοπίου. Ε, βγάλουμε δηλαδή το στοιχείο της περιπλοκότητας και επιτρέψουμε με ευχαριστήρο τρόπο μπορεί ο, Χρήστ, ο Γεωργός να το χρησιμοποιήσει το μέσο αυτό. Αλλά όπως είπα, η κατεξόδηση ε, πράξη για την οικολογικοποίηση είναι σε διαδικασία επισκόπησης τώρα και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την ευκαιρία να τη στις λεπτομέρειες της αργότερα. Την έχουμε συστήσει μαζί σας. Αλλά θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε για να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της πράξης και θα σταματήσω. Το ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθύντα. Ο κύριος Ντές έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θέλω εδώ να επισημάνω κάτι στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή να μας κάνει αναλυτική κατάθεση των κατεξιοδότηση πράξεων. Αυτές οι 14 όμως τους κατεξιοδότηση πράξεις, ο κύριος Χόγκαν και η Επιτροπή ολόκληρη δεν φάνηκαν ετεθειμένοι να μας τις παρουσιάσουν αναλυτικά. Όταν υπάρχουν 14 νομοθετήματα που μέσα σε μία κατεξιοδότηση πράξη καλύπτονται, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ξανακοιτάξει την κατάσταση. Ας μην ε, επιμείνει σε αυτό, γιατί βεβαίω δεν θα δεχθούμε περιορισμό των ε, εξουσιών του Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου. Επίσης με συγκλονίζει η απάντηση σε σχέση με τα φυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα. Μάλλον δεν έχετε ιδέα για το τι γίνεται σε σχέση με τις καλλιέργειες. Έχω βαρεθεί πια να έρχονται οι διάφοροι υπάλληλοι και να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε χωρίς να έχουν ιδέα για το τι στην πραγματικότητα συμβαίνει και συγγνώμη που μίλησα τόσο μα τόσο απερίφραστα. Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό, ούτως όλους πολύ σύντομα. Αλμπέρ, έχεις Εσύ που είσαι σε διαρκή επαφή με τον ε, Γεωργό, με την πραγματικότητα της Γεωργίας και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να φτάσουμε σε αυτή την απλοποίηση και την οικολογικοποίηση. Και πρέπει αυτό να το καταστήσουμε ορατό με τις δράσεις μας, με αποφασιστικότητα βεβαίως, την οποία διαγιγνώσκω στη δική σας στάση, η οποία αποφασιστικότητα μας λέει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την οικολογικοποίηση και την απλούστευση. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δοθέσατε. Θα επανέλθουμε, όπως είπα, το ταχύτερο. και σημειώνουμε βεβαίως τις ε, παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων. Επισημένω πως πρόκειται για παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώνονται πάνω απ' όλα στο όνομα των γεωργών. Οι γεωργοί βλέπουν τα πράγματα έτσι. Το είπατε κι εσείς. Και όλοι ε, θέλουμε οι αλλαγές που προτείνουμε να βαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και να είναι επωφελής για τους Γιώργους. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της θέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, γεωργικές διακλαδικές οργανώσεις. Έγιναν ε, μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση της κατάστασης των διακλαδικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρόκειται για μια ε, πρώτα ανάλυση των περίπλοκων εθνικών διατάξεων που διέπουν τις διακλαδικές διακλαδικές οργανώσεις και η ανάλυση που γίνεται ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για το ρόλο τους στην ε, αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα και αναλύει τη λειτουργία, τα ωφέλη και τις προκλήσεις των διακλαδικών οργανώσεων. Εμείς θέλουμε φυσικά να ενισχύσουμε τη θέση του γεωργού στην αλυσίδα προμήθειας ε, των τροφίμων και στην αλυσίδα και να ενισχύσουμε και τη διαπραγματευτική του ισχύ και τα εισοδήματά του. Και θα δούμε αν συμβάλλουν στο στόχο αυτό οι διακλαδικές οργανώσεις. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη, η κυρία Κλίμαν, που θα μας κάνει αυτή την νομική ανάλυση των διακλαδικών οργανώσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις διακλαδικές ε, οργανώσεις ε, των αγαπητών ε, που ρυθμίζονται στον κανονισμό της κοινή αγοράς. Όπως λέει ο πρόεδρος, σωστά μπορούν να έχουν σημαντικές αρμοδιότητες, αλλά πριν να περάσουμε στην ίδια τη μελέτη που έγινε από την Arcadia International και το Πανεπιστήμιο του Βάχενιγεν, θα ήθελα για λίγο να σας υπενθυμίσω το τι είναι ακριβώς αυτές οι διακλαδικές οργανώσεις. Ε, θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο αυτορύθμισης και ενώ οι γεωργικές. Η έκθεση του Ιανουαρίου φέτος από μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών μίλησε πάρα πολύ για τη συλλογική δράση των γεωργών σε σχέση με τις, παραγω... με τις οργανώσεις παραγωγών. Βρίσκουμε ελάχιστα για τις διακλαδικές οργανώσεις ε, και γιατί αυτό. Θεωρώ πως ένας λόγος είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε του ποιες συγκεκριμένες οργανώσεις έχουμε στο πλαίσιο των διακλαδικών οργανώσεων, τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, για την πρώτη διαφάνεια, πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε ότι είναι κάθετες οργανώσεις, όπως ρυθμίζονται δηλαδή στον κοινό κανονισμό αγοράς. Αυτό το οποίο βλέπουμε εκεί πέρα είναι ακριβώς η εκπροσώπηση των παραγωγών συν του τομέα της μεταποίησης ή και της λιανικής. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ότι οι περισσότερες διακλαδικές οργανώσεις είναι ε, οι λεγόμενες ε, βραχίες τέτοιες οργανώσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι περιλαμβάνουν μόνο το τομέα της παραγωγής και της μεταποίησης από τις 123 τέτοιες αναγνωρισμένες οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 18 περιλαμβάνουν και τον τομέα της λιανικής πώλησης. Όμως η μελέτη δημιούργησε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε το εργαστήριο στις 23 Μαρτίου και είδαμε πως πολλές από τις οργανώσεις Λιανικής ε, εγγράφησαν και ζήτησαν συμμετοχή στο συνέδριο. Πρέπει όμως να τονίσουμε και να απαντήσουμε το ερώτημα του Κοινοβουλίου. Το ποιος είναι ο ρόλος δηλαδή. Το τι ε, μπορούν και το τι δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι οργανώσεις. Και σαφώς ο ε, κανονισμός κοινής αγοράς λέει ότι δεν μπορούν να έχουν εμπορικές δραστηριότητες, ότι δεν θα μεταποιήσουν, δεν θα παραγούν αυτό, ζητάει ο κανονισμός κοινή αγοράς και είναι κατανοητό γιατί από πλευράς ε, ε, δικαίου του ανταγωνισμού, εάν υπάρχει ολόκληρη η αλυσίδα της ε, παραγωγής χωρίς τον καταναλωτή είναι περίπλοκα τα πράγματα, ειδικά εάν ταυτόχρονα παράγει και μεταποιεί κανείς. Λοιπόν, διαφέρουν οι οργανώσεις αυτές από τις οργανώσεις παραγωγών, να βλέπουμε ότι είναι μια πλατφόρμα διαλόγου, έρευνας, βοηθούν στο να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές και κυρίως το ότι είναι συνομιλητές των κρατών μελών, αλλά επίσης θέλουν να μιλήσουν και με εμάς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν βεβαίως πολύ καιρό πριν από τον κανονισμό του 2013 στον τομέα των ε, τροφίμων ε, και των οπωροκυπευτικών, αλλά το 2013 πλέον οι κανόνες έγιναν οριζόντιοι. Τώρα η μελέτη τα εξετάζει όλα αυτά, όπως είπατε σωστά, το τι συμβαίνει. Η μελέτη λοιπόν ερεύνησε το τι εθνική νομοθεσία υπάρχει για τις διακλαδικές αυτές οργανώσεις, το τι συμβαίνει, ποιος υπάρχει, σε ποια κρατημέλη, σε ποιον κλάδο, το τι κάνουν και τρίτον Ποια είναι τα ωφέλη που ε, μπορούν να έχουν για τους γεωργούς ε, ή μπορούν να έχουν ωφέλη μόνο για τους γεωργούς ή για ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα και ποιους όρους ε, χρειάζονται οπωσδήποτε για να μπορούν να λειτουργούν. Προφανώς ένας μεγάλος παράγων είναι η χρηματοδότηση. Πηγαίνοντας λοιπόν στην εθνική νομοθεσία. Θα το περάσω αυτό πάρα πολύ γρήγορα γιατί ούτως ή άλλως ισχύει απευθείας ο κανονισμός. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε ότι ε, το κράτος μέλος το οποίο είχε από το 1975 την παλαιότερη παράδοση τέτοιων οργανώσεων είναι η Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία τότε υπήρχαν κάθετοι διακλαδικοί οργανισμοί, αλλά είχαν δημόσια φύση. Σήμερα είναι ιδιωτικοί οργανισμοί. Έχουμε δύο-τρεις τέτοιες μόνες ε, οργανώσεις στην Γαλλία όπου εκπροσωπείται το κράτος, αλλά κατά κανόνα είναι ιδιωτικές οργανώσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν κάνει η Εθνική Νομοθεσία είναι να ορίζει κανόνες για την αναγνώριση για επέκταση κανόνων και βεβαίως για τα τέλη. Εν ολίγης, είναι μια υπόθεση κρατών μελών, αλλά τι σημασία έχει αναγνώριση. Κοιτάξτε, ο κανονισμός οργάνωσης της αγοράς εξαιρεί τους, κανονισμού, τους οργανισμούς αυτούς από την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού εάν είναι αναγνωρισμένοι ως ένα βαθμό. Θα θυμάστε όμως αυτά τα οποία σας είπα πριν ότι δεν θα παράγουν, δεν θα μεταποιούν. Υπάρχει και άλλη μια έντολη που λέει δεν θα μοιράζεται τις αγορές, δεν θα καθορίζεται τις τιμές και δεν θα ορίζεται Οπότε οι διακλαδικέ οργανώσει λειτουργούν πάρα πολύ καλά, αλλά εντό συγκεκριμένου πλαισίου και το πλαίσιο αυτό ορίζεται και από του κανόνε του ανταγωνισμού. Η επέκταση των κανόνων είναι κάτι το ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον μέρος της, ε, μέρος της ε, δουλειάς των οργανισμών αυτών, όπως επίσης και τα τέλη. Σύμφωνα με τις δυνατότητες επέκτασης των κανόνων, ένας τέτοιος διακλαδικός οργανισμός μπορεί παραδείγματος χάρη να αναπτύξει μία προδιαγραφή, π.χ. το μέγεθος ενός πεπονιού και μπορεί μετά να πάει στο κράτος μέλος και το κράτος μέλος να επεκτείνει αυτή τη συμφωνία σε μη μέλη. Δηλαδή ακόμα και άτομα τα οποία δεν εκπροσωπούνται στην διακλαδική οργάνωση πρέπει μετά να εφαρμόζουν τους κανόνες της διακλαδικής οργάνωσης. Και για την επιβολή τελών αυτό είναι ακόμη πιο εκπληκτικό. Δηλαδή μπορεί ε, σε πληρώνουν προφανώς τα μέλη σου, αλλά εάν θεωρείς ότι κάνεις ε, καλό στον κλάδο συνολικά, μπορείς να απευθυνθείς στο κράτος, εάν έχει μια ανάλογη πρόβλεψη που δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη, και να ζητήσεις βασικά ακόμα ε, και όσοι δεν είναι μέλη σου να σε πληρώνουν. Βλέπετε ότι μόλις 19 κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει σχετική νομοθεσία Και μετά θα δείτε στην επόμενη διαφανεία από τα 19 μόνο 8 κράτη-μέλη έχουν όντως αναγνωρίσει τέτοιους οργανισμούς. Οπότε θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη ε, μη εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Βλέπετε τα κρατημέλη, η Γαλλία με τη μεγαλύτερη παράδοση, αλλά και η Ισπανία με 63 τέτοιες οργανώσεις διακλαδικές που υπάρχουν σήμερα σήμερα τον Ιούνιο του 2016 που έγινε η μελέτη αλλά και στην Ουγγαρία, την Ιταλία, τρεις στην Ολλανδία, πέντε στη Ρουμανία και 4 πέντε στην Πορτογαλία. Ε, γιατί λέμε 119 ε, συν 4 ε, στην Γαλλία Κάποιες τέτοιες οργανώσεις έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες γιατί προϊόντα που αφορούν το κονιάκ και τα σαλιγκάρια δεν είναι γεωργικά προϊόντα υπό την έννοια του κανονισμού. Λοιπόν, πού βρίσκονται, πού δραστηριοποιούνται αυτοί οι οργανισμοί, κυρίως στο εθνικό επίπεδο, κάποιος στο περιφερειακό επίπεδο, κυρίως στον τομέα του ίνου και τροφίμων και οπορεκπαιδευτικών και στον τομέα των γαλακτοκομικών. Λοιπόν, έκτοτε είχαμε την πρώτη τέτοια οργάνωση ευρωπαϊκή ε, για τον καπνό που αναγνωρίστηκε από την Ιταλία και η Γερμανία η οποία μέχρι στιγμής δεν είχε δει το θέμα ζεστά μόλις αναγνώρισε την πρώτη τέτοια οργάνωση στον τομέα της ζάχαρης. Και παρενθετικά Ιστορικά οι διακλαδικές οργανώσεις ε, σχηματιζόταν γιατί η αλυσίδα ε, έβλεπε ότι υπάρχει μια κρίση, δηλαδή ήταν συνήθως σε μια κρίση, αλλά αν ρωτήσουμε τώρα παραδείγματος χάρη τον εκπρόσωπο της γερμανικής οργάνωσης ε, για την ζάχαρη, γιατί το κάνετε αυτό, ήταν γιατί είπαν ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την εξαίρεση από τους κανόνες του ανταγωνισμού και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ε, για να δείτε βασικά το τι ε, σημαίνει διακλαδική οργάνωση. Το θέμα είναι χρηματικό. Βλέπουμε στην Ισπανία όταν σταμάτησε η χρηματοδότηση του κράτους ουσιαστικά επέκτηναν την χρηματοδότηση μέσω την επιβολή, της, ε, επιβολής τελών κάτι το οποίο οι Γάλλοι λένε υποχρεωτικά εθελοντικά τέλη. Μια ενδιαφέρουσα διατύπωση. Στη Ρουμανία βλέπουμε πως ε, έχουν έναν προπολογισμό κάτω από 10.000 ευρώ. Στη Γαλλία υπάρχουν οργανώσεις που έχουν προπολογισμό πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε υπάρχουν και διαφορετικές ε, παραδόσεις στη Γαλλία. Δηλαδή είναι συνηθισμένοι στο να έχουν μεγάλες οργανώσει που τους εκπροσωπούν σε άλλα κράτη-μέλη μόλις ξεκινούν. Αλλά όταν μιλάμε εμεί μαζί του και αυτό το επιβεβαίωσε και η μελέτη, κάποια ε, χρηματοδότηση για να μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν. Λοιπόν, οι στόχοι του ε, ανέφερα πολλές τέτοιες οργανώσεις ε, ερωτήθησαν, δηλαδή ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι στόχοι σας να ε, θεωρούν ότι πρέπει να είναι μια πλατφόρμα για να συνεννοούνται οι διάφοροι κατά καθόλου το μήκος της αλυσίδας. Οπότε το όφελος ε, μοιράζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα και τελικά ελπίζουμε και στους γεωργούς. Επίσης, το να αναπτύσσουν υποδείγματα συμβάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τους συναλλασσόμενους. Και τώρα πια κάνουν και έρευνα. Έρευνα για το προϊόν, κάτι το οποίο ωφελεί τους πάντες. Όχι για ένα συγκεκριμένο τμήμα της αλυσίδα για το προϊόν. Και βεβαίως είναι και συνομιλητές κρατικών φορέων και αυτό είναι κάτι το οποίο αρέσει στα κράτη, γιατί αν θέλουν έναν κλαδικό κανονισμό και έχει μία φωνή ο κλάδος, ε, είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον και αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχω πει και ζητώ συγγνώμη, ε, είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σε κάποια κράτη μέλη, σε 6-7 Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, είναι ότι λένε εγώ θέλω με έναν οργανισμό να μιλάω ανά ή κατηγορία ή κλάδο. Οπότε χ κλάδε θέλω να κάνετε μια οργάνωση. Οπότε, γιατί δεν έχουν νομοθετήσει κάποια κράτη-μέλη ποτέ και δεν έχουν αναγνωρίσει διακλαδική οργάνωση. Αυτό το οποίο θέλαμε να, και εσείς θέλατε να δείτε με αυτή την μελέτη, είναι να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια φιλοδοξία να νομοθετήσουμε. Όχι, θέλαμε απλά να δούμε το τι συμβαίνει. Και δεν είναι αυτόματο το ότι πρέπει να συσταθεί μια διακλαδική οργάνωση αν υπάρχουν άλλα μέσα και λειτουργούν. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης από πού θα ξεκινήσουν. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να βοηθήσουν γιατί μπορεί να μην ξέρουν. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο για μια οργάνωση και σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μια δυσπιστία όσον αφορά την κάθε συνεργασία. Αλλά επίσης ε, έχουμε πάει και στην Κροατία που υπάρχει μια αργή ε, υιοθέτηση των ε, οργανώσεων παραγωγών. Οπότε αν δεν έχουν οργανωθεί ούτε καν η παραγωγή, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθετοποιημένη οργάνωση γιατί οι διακλαδικές ε, οργανώσεις έχουν ως εξής 75 έως 80% του πρωτογενούς τομέα εκπροσωπείται στις διακλαδικές οργανώσεις δηλαδή η παραγωγή έχουν λόγο ε, στι διακλαδικές οργανώσεις. Αλλά αν δεν είναι αυτοί οργανωμένοι δεν θα υπάρξει βεβαίως και διακλαδική οργάνωση. Και μετά, εντάξει, αυτό ίσως φαίνεται αντιφατικό αλλά δεν είναι, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ήδη μεγάλες καθετοποιημένες οργανώσεις όπως στην Γερμανία παραδείγματος χάρη όπου υπάρχουν ισχυροί συνεταιρισμοί και για τον λόγο αυτό δεν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη στο να πάνε στην αναγνώριση διακλαδικών οργανώσεων και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε πως ε, επηρεάζεται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας οργάνωσης. Είπα εισόδημα, ενημέρωση αλλά και το μέγεθος. Λέμε πως ε, ε, σε πολλά κατημέλια αρέσει το μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά μεγάλο μέγεθος μπορεί να κάνει την δουλειά τους εσωτερικά πιο δύσκολη, γιατί ένα είναι το κοινό έβριμα της μελέτης, το οποίο είναι ότι σε μια διακλαδική οργάνωση ε, δουλεύουν συνενετικά. Μπορούν να ψηφίσουν, αλλά δεν το κάνουν, γιατί αν είναι να ψηφίσουν, σημαίνει πως ε, δεν συμφωνούν. Οπότε τι συμφωνία θα έχουν, δηλαδή, αν είναι να ε, ψηφίσουν ε, ενάντια στη θέληση των μεταποιητών ή των παραγωγών. Και μας λένε όλοι ότι δουλεύουμε με την συνένεση και ξέρουμε βεβαίως πως όταν είναι και λίγοι ε, γίνεται καλύτερα αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρουν το τι πρέπει να κάνουν θέμα εσωτερικής οργάνωσης και το τι μπορούν να κάνουν. Πρέπει δηλαδή να είναι σαφής η κανόνες και η ρυθμιστική και του ανταγωνισμού και η σχέση επίσης με τις αρχές είναι πολύ σημαντική. Στη Γαλλία όπου υπάρχει χρόνια το σύστημα υπήρχαν συχνές επαφές και για πρωτοβουλίες, για επέκταση κανόνων, για επέκταση τελών και αυτό βοηθάει να λειτουργεί καλύτερα η αλυσίδα και οι διακλατικές οργανώσεις. Αλλά θεωρούμε ότι, έχοντας διαβάσει τη μελέτη, είναι ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η διαφάνεια. Ειδικά αν θέλουμε να πληρώνουν και τα μη μέλη, αν θέλουμε τα μη μέλη να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές, π.χ. το μέγεθος ενός πεπονιού, το οποίο αποφάσισε ένας οργανισμός τον οποίο δεν είμαι μέλος, χρειάζεται διαφάνεια. Αυτό προέκυψε από τη μελέτη, αλλιώς και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω Ποιο είναι το όφελος ε, ενό διακλαδικού οργανισμού. Ναι, είναι καλό υπό όρους, αν ξέρει το τι κάνει, αν μιλάει με μια φωνή και αν ε, έχει ως ε, συνομιλητή τις αρχές που αντιλαμβάνονται τους κανόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση της έκθεσης. Ενδιαφέρουσα, σημαντική και σας ευχαριστούμε για την πυγμή, την αποφασιστικότητα με την οποία παρουσιάσετε την έκθεσή σας και που δείχνει τη δέσμευσή σας. Γι' αυτό και ήταν πολύ πιστική η παρουσίαση χάρη σε αυτή την αποφασιστικότητα. Ο λόγος τώρα στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Ο κύριος Νταντάν πρώτα, που είναι και εμπειρογνώμονας για αυτά τα θέματα των αγορών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας παρουσίασε τη σχετική μελέτη. Την ευχαριστώ και για τον ενθουσιασμό της βέβαια, αλλά και για την εκπόνηση αυτής της μελέτης που δείχνει τις ευκαιρίες ε, που προκύπτουν από τις ε, διακλαδικές οργανώσεις. Το 2013 συστήσαμε ένα, μια εργαλειοθήκη. Εναπόκειται τους διάφορους φορείς να αξιοποιήσουν τα επιμέρους εργαλεία αυτής της εργαλειοθήκης, να δουν ποια είναι τα πιο κατάλληλα, ανάλογα με την εθνική τους κατάσταση. Και ίσως δεν είναι αρκετά γνωστά αυτά τα εργαλεία. Οπότε η έκκλησή μου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ίσω και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσουμε μια πιο δυναμική πολιτική για να προβάλλουμε αυτά τα εργαλεία ρυθμίσης των αγορών. Γιατί τέτοιου εργαλεία μπορούν να προλάβουν τις κρίσεις, να συμβάλλουν στη διαχείριση των κρίσεων και να αποτρέψουν και κάποιες κρίσεις ίσως. Θα σας αναφέρω ένα γαλλικό παράδειγμα που είναι ενδεικτικό. Η σαμπάνια για παράδειγμα. Μία διακλαδική οργάνωση ε, διαχειρίζεται τη σαμπάνια. Από το 1941 χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο της διακλαδικής οργάνωσης και χάρη σε αυτή τη διακλαδική οργάνωση έκανε η σαμπάνια το ποιοτικό άλμα της ε, ε, και κέρδισε τη δημοτικότητα, τη φήμη και τη διεθνή προστασία που έχει σήμερα. Και στην Ιταλία ή την Ισπανία επίσης έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα διακλαδικών οργανώσεων για φρούτα για παράδειγμα που είναι ε, παραδείγματα προς μίμηση για τη διαχείριση της αγοράς και επιτρέπει όλο τον κλάδο να κάνει ένα βήμα προόδου και σε τεχνικό επίπεδο, αν το επιτρέπει η έρευνα, αλλά και σε επίπεδο γνώσης της αγοράς, προσαρμογής της αγοράς στις ανάγκες του καταναλωτή, διαχείριση των κρίσεων, αλλά φυσικά χρειάζεται διαφάνεια. Γιατί πρόκειται για ένα εργαλείο, όχι για πανάκια. Και ο καθένας θα πρέπει να το αξιοποιεί και να το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν γνωστή σαμπάνια επειδή ήταν καλή. Mm. Απλώς. Ο κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πολύ ενημερωτική παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την αναγνώριση τέτοιων οργανώσεων. Μια στιγμή. Συνεχίστε. Θα ήθελα λοιπόν να ε, θέσω κάτι συγκεκριμένο ε, το οποίο αφορά την αναγνώριση τέτοιων οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή οι διακλαδικές οργανώσεις μπορούν να ε, συσταθούν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 1 και παράδειγμα 1 του κανονισμού. Το πρόβλημα είναι ότι η κατάταξη των προϊόντων στο παράρτημα δεν είναι ε, τελείως λογική σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα, στον τομέα της γεωργίας, στην χώρα μου, στην Ολλανδία, υπάρχει ένας ε, οργανισμός ο οποίος ε, προσπάθησε να συσταθεί στον τομέα ακριβώς της αεροτρέας γεωργίας. Όμως θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικά για τις πατάτες ξεχωριστοί οργανισμοί πριν προχωρήσουν ε, σε σύσταση ενός οργανισμού ο οποίος ε, παραδείγματο χάρη θα εκπροσωπούσε και άλλες ε, καλλιέργειες π.χ. τον καφέ ή οτιδήποτε άλλο σε έναν διακλαδικό οργανισμό. Το πρώτο μου λοιπόν ερώτημα είναι θεωρείτε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στην παρέμβαση και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ε, εδώ πέρα. Εντάξει, καλή η παρουσίαση, αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα όσον αφορά την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Η κυρία Ράνς Καρσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση και να ε, συμμεριστώ τον ενθουσιασμό της για το ρόλο των διακλαδικών οργανώσεων στην αλυσίδα τροφίμων ε, την άποψή της και είμαι υπέρμαχος των διακλαδικών οργανώσεων. Εμείς από το 1994 έχουμε νόμο που ρυθμίζει τις διακλαδικές οργανώσεις ε, στο ελαιόλαδο, στο, στον ίνο, στις επιτραπέζιες ελιές, στις πατάτες. Επίση έχουμε διακλαδική οργάνωση του κρασιού της Ριόχα που βοήθησε ιδιαίτερα στην οργάνωση του κλάδου και διευκόλυνε την ε, σύναψη συμφωνιών και την αποτροπή συγκρούσεων την τελευταία δεκαετία. Και είμαστε κατενθουσιασμένοι με τη διακλαδική οργάνωση τη Ριόχα. Θέλουμε λοιπόν ε, να προωθηθεί ο ρόλος των διακλαδικών οργανώσεων και να ενισχυθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λέτε ότι ισχυροί συνεταιρισμοί παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των διακλαδικών οργανώσεων, γιατί εγώ έχω την αντίθετη ε, εντύπωση από την πείρα μου. Εγώ θεωρώ ότι και οι καλά οργανωμένοι συνεταιρισμοί οικειοθελώς ε, συμμετέχουν και είναι και ιδιαίτερα δραστήριες, ε, δραστήριες στις διακλαδικές οργανώσεις. Γιατί λοιπόν τις θεωρεί εμπόδιο, τους θεωρεί εμπόδιο τους συνεταιρισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα να δώσουμε ε, περισσότερη φωνή σε αυτέ τι διακλαδικέ οργανώσει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκή πολιτική και στη λήψη αποφάσεων, γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ευέλικτο και απαραίτητο στην τροφική αλυσίδα. Εμεί ε, θέλουμε να αναγνωριστεί ο ρόλος του στην τροφική αλυσίδα και φυσικά να ρυθμιστεί. Και η, ε, η ισπανική επιτυχία θα μπορούσε να είναι παράδειγμα προς μίμηση όπως και η γαλλική επιτυχία, το γαλλικό παράδειγμα. Φυσικά ως ε, Επιτροπή Γεωργίας πραγματοποιήσαμε αποστολή στη Ριόχα και πραγματικά είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα και υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση. Κύριε Ντελάη, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που ανέλαβε να παρουσιάσει το θέμα αυτό. Πρόκειται για έναν από τους άξινες, υπενθυμίζω, της ε, έκθεσης για την πληθυκότητα, για την καταπολέμηση δηλαδή, της των τιμών στα ιωρικά προϊόντα που θέτησαμε πέρσι με μόνο βέβαια ψόγο ότι έγινε αυτή η παρουσίαση Παρασκευή και δεν είχαμε παρουσία πολλών βουλευτών και εγώ ήδη θα είχα πολλά να, να ε, επισημάνω. Είπατε για τη Γαλλία ότι έχουμε μακρά παράδοση. Ναι, αλλά έχουμε και διάφορους ε, τύπους διατομεακών ε, οργάνων εγώ ήμουν για πολλά χρόνια σε έναν οργανισμό διατομιακό Λαχανικών και έναν άλλον που είχε περισσότερο οικονομική στόχευση και αυτοί περισσότερο με ενδιαφέρουν. Γιατί εγγύησε ότι θα υπάρχει ένας τόπος, μια πλατφόρμα που όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διανομή της αλυσίδας των τροφίμων, τροφίμων ο παραγωγός, ο μεταποιητής, ο χονδρέμπορος, ο μεταφορέας, ε, ακόμη και ο, οι ο Λιανικής, θα μπορούν σε αυτήν την πλατφόρμα να συζητούν, να καταλήγουν και σε συμφωνίες για την ποιότητα των προϊόντων και έτσι να εξασφαλίσουν μια καλή αλυσίδα τροφίμων. Πρέπει να ενθαρρυνθούν και είναι ο ρόλος της αυτός οι οικονομικοί φορεί να αναπτύξουν τέτοιου είδου διατομιακού ε, φορεί. σε μια αλυσίδα για μένα όσο δυνατόν μακρότερη, μακρύτερη γιατί βέβαια η γεωργία μόνη τη χωρί το εμπόριο δεν μπορεί να δώσει απαντήσει και χάρη στην αλυσίδα αυτή μπορούμε να έχουμε στο δυνατόν καλύτερη αλυσίδα. Ο κύριο Ανδρίου, πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ θέλω να Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πολύ καλή δουλειά της. Στην ίδια γραμμή με τα όσα ακούστηκαν πριν από τους συναδέλφους. Το ζήτημα βέβαια, το κύριο είναι το εισόδημα, η προσθέμενη αξία αυτών των τετομεακών οργανώσεων και η αριστεία που μπορούν να εξασφαλίσουν και με την ψηφοφορία για τον κανονισμό Omnibus που αναφέρθηκε νωρίτερα. Νομίζω ότι έρχεται ακριβώς σε έφθετη στιγμή, γιατί θα το ψηφίσουμε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επαγρυπνούμε προς τα όρια των οργανώσεων. Ανέφερε η κυρία Ντελάη ότι υπάρχει και η παραγωγή, η μεταποίηση, μεταφορά, ε, η διανομή. Υπάρχουν διάφορα τμήματα και πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερα ως προς την κατανομή των εσόδων προς όφελος των παραγωγών. Γιατί το να υπάρχει αυτή η οργάνωση δεν μας απαλλάσσει από τον έλεγχο του ανταγωνισμού. Και ε, λέω ότι βεβαίως καλό είναι αυτό να γίνεται οπωσδήποτε προκαταβολικά και όχι εκ των υστέρων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και αυτό το λέω και τι πιστεύω ότι περισσότερο παρά ποτέ είναι απαραίτητες οι διατομεακές οργανώσεις για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ, Αγγουιλέρα. Ευχαριστώ. Με χαροποιεί αυτή η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διακλαδικές οργανώσεις. Και δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι που τα περισσότερα μέλη που μείναμε τουλάχιστον αυτή τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι Γάλλοι και Ισπανοί. Γιατί ε, είχαμε πολύ θετική εμπειρία πρώτα στη Γαλλία που έχει και πιο μακροχρόνια πείρα και μετά στην Ισπανία από τις διακλαδικές οργανώσεις. Δεν ξέρω γιατί στις υπόλοιπες χώρες δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένη εφαρμογή. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε και να προσθεριστούμε τα κράτη-μέλη σε αυτή την προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι οι διακλαδικές οργανώσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και σίγουρα στην πατρίδα μου, όπως είπε η κυρία Ερά, στην Ισπανία, έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας. Δεν είναι πανάκια βέβαια, δεν είναι θαυματουργή λύση, αλλά ως μέσο εργαλείο ρύθμιση της αγοράς είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος τους. Θα ήθελα τώρα να αξιοποιήσουμε τη δική σας πείρα και να δούμε ε, αν θα ήταν χρήσιμο να περιλάβουμε τις διακλαδικές οργανώσεις και τη διανομή. Να έχουμε όλη την έκταση δηλαδή, της αλυσίδας από την παραγωγή, την ε, εμπορία του τους εμπόρους χονδρικής, λιανικής και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τη διανομή. Δεν ξέρω αν τα σούπερ μάρκετ θα, θα ήθελα να συμπεριληφθούν, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η εκπροσώπηση στις εκλατικές οργανώσεις, τόσο μεγαλύτερη η ισχύ τους. Να ενισχύσουμε πάντως τις οργανώσεις και ίσως να ενισχύσουμε και την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί... Ε, μια και είναι μοναδικό το ευρωπαϊκό εμπόριο, χρειαζόμαστε πιο εκτεταμένη νομοθεσία που να καλύπτει και τις διακλαδικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ. Οφείλω να ομολογήσω ότι για πρώτη φορά ήταν τι διακλαδικέ οργανώσει όταν ασχοληθήκαμε με το γαλακτοκομικό τομέα, τη δέσμη μέτρων. Και ο κύριος Νταντά έχει δίκιο ότι σε μερικέ χώρες είναι πολύ πιο γνωστές αυτές οι οργανώσεις. Τότε κάναμε διεξοδική έρευνα και στη πατρίδα μου δεν βρήκαμε σχεδόν τίποτα. Πάντως στη Γαλλία και την Ισπανία είναι πολύ σημαντική η παρουσία του και φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ευρέως οι διακλαδικές οργανώσεις ως εργαλείο στις δύο αυτές χώρες. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, οι διακλαδικές οργανώσεις έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις χώρες του Νότου από τις χώρες του Βορρά. Υπάρχει μια διαφορά Βορρά-Νότου, ένα χάσμα Βορρά-Νότου ή είναι θέμα ενδιαφέροντος των κρατών μέλων ε, μερικά κράτη-μέλη το θεωρούν χρησιμότερο εργαλείο και πιο ε, αποτελεσματικό. Επίσης, ε, με, άκουσα με ενδιαφέρον αυτά που είπατε για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι διακλαδικές οργανώσεις είναι αντίπαλοι των συνεταιρισμών, αν και ίσως σε μερικές χώρες αυτή η εντύπωση υπάρχει. Και ανακύπτω ερώτημα, μήπω υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ διακλαδικών οργανώσεων και συνεταιρισμών. Έτσι θα εξηγούνταν οι απροθυμία μερικών κρατών μελών να τι ενισχύσουν. Από ό,τι ακούσαμε σε μερικές περιοχές, όπως στην ε, Γαλλία για τη σαμπάνια και στην Ισπανία με το κρασί της Ριόχα, η δράση τους ήταν αποτελεσματική και ίσως από αυτά τα παραδείγματα θα πρέπει να διδαχθούμε και σε άλλες περιφέρειες και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αγορητών και θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον, στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σχολιάσει μεταξύ άλλων και αυτά που είπα ο κύριος Νίκολσον. Για μερικούς ε, κλάδους, για μερικούς τομείς, οι διακλαδικές οργανώσεις είναι πολύ καλό εργαλείο και συμπληρώνουν ε, ίσως την αγορά. Μήπως όμως έρχονται σε ανταγωνισμό με άλλες οργανώσεις σε ορισμένες αγορές. Θα ήθελα για αυτό το θέμα του ανταγωνισμού των διακλαδικών οργανώσεων με άλλες οργανώσεις ε, να μας μιλήσετε πιο εκτενώς. κυρία Κίλιμαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα πολύ σημαντικές ε, ερωτήσεις. Βεβαίως, ε, ρώτησε ο κύριος Δοντέ αν θα πρέπει να προβεί σε μια συνειδητή απόφαση το κράτος μέλος και αν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Ε, περί αυτού ακριβώς πρόκειται, αυτό λέει και η μελέτη μας, το χρησιμοποιείτε και το λέμε ρητά όπως σας ε, βολεύει, όπως ε, ταιριάζει τις ανάγκες σας. Ε, είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα μοντέλο κράτους μέλους στα λοιπά κράτη-μέλη. Γιατί βεβαίως Μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση για ένα κράτο που έχει διατομεακή οργάνωση εδώ και 40 χρόνια και ένα άλλο που δεν έχει. Άρα το βασικό είναι η ιδέα του διατομεακού δεσμού. Δεν αποφασίζει ο δεσμός αν θα υπάρχει, αλλά εξετάζεται αν μπορούν να μπουν άλλοι φορείς που δεν ανέχουν σε αυτόν και πάνω απ' όλα αν εξυπηρετεί το ίδιο το κράτος μέλος. Αυτό για να υπογραμμίσω πάνω απ' όλα ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Έχει μεγάλο, μεγάλη σημασία αυτό. Αναφερθήκατε στη Γαλλία, τη Σαμπάνια. Πολύ σημαντικό βεβαίως. Και έχουν ε, πολύ συχνά επισημένο οι διατομιακοί φορείς ε, συσταθεί σε περίοδους κρίσεως, αλλά, για να δώσω και το παράδειγμα του τομέα της ζάχαρης ε, στη Γερμανία, έχουν αξιοποιηθεί ε, ως εργαλεία πολύ χρήσιμα και σε περίπτωση κρίσεως και το άρθρο 222, με εξαίρεση βεβαίως την κρίση το Καλακτοκομικό έχει ιδιαίτερη, ιδιαίτερα βοηθήσει και ο σχετικός κλάδος της Ζάχαρη στη Γερμανία μας είπε εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε να οργανωθούμε αφού εμφανιστεί η κρίση. Εμείς πρέπει να οργανωθούμε πριν εμφανιστεί η κρίση. Άρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τομεακό ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλήματα κρίσεως. Αλλά ο καθένας τα κρίνει βέβαια. Τώρα τι σημαίνει ότι η παρατήρηση ότι δεν είναι λογικός αυτός ο κανονισμός. Ε, προφανώς δεν είναι για μένα, ε, δεν είναι δικό μου καθήκον ως εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλήσω για το αν είναι λογικός ή όχι ένας ε, κανονισμός που αναφέρεται πραγματικά, στην κοινή οργάνωση αγοράς. Πολλές φορές μπορεί να προκύπτει πρόβλημα όταν ένα προϊόν μπαίνει σε ένα τομέα μαζί με ένα άλλο. Από την άλλη μπορούμε να δούμε και διαφορετικά την κατάταξη με τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και το γιαούρτι που χωρίς ζάχαρη μπορεί να θεωρηθεί μη γεωργικό προϊόν, ενώ μαζί με ένα άλλο προϊόν μπορεί να μπει στην κατηγορία των γεωργικών προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει, οι περιορισμοί είναι νομικοί, καθαρά νομικοί περιορισμοί και το έχουμε επισημάνει βέβαια όταν τα κρατημέλη μας ρώτησαν ε, αν υπάρχει κάποια διέξοδος. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε διασταλτική ερμηνεία. Είναι σε οι κανόνες για ένα γεωργικό κλάδο, αλλά δεν θέλω να ε, επισέλθω σε μια αξιολόγηση ποιοτική. Η άλλη ερώτηση για τη Ριόχα της Ισπανίας. Είπα έτσι ώστε να μην ήταν σαφής οι παρατηρήσεις μας. Γιατί να αποτελούν πρόβλημα οι εθνικές διατάξεις. Ε, αυτό σε συνδυασμό και μετά όσο είπε και ο κύριος Νίκολσον, ε, έχει ως απάντηση τον ανταγωνισμό μεταξύ συνεταιρισμών και διατομεακών δεσμών. Μπορεί να υπάρχουν και τα δύο φυσικά. Αλλά με διαφορετικέ λειτουργίες ίσω. Εάν εφαρμόσουμε δηλαδή, τον ορισμό του συνεταιρισμού, όπως τον είδαμε στην μελέτη του 2012, ο συνεταιρισμός δηλαδή είναι μια οντότητα που έχει ε, που ε, υπόκειται στον έλεγχο του χρήστη και διαμορφώνεται με βάση την πούληση του χρήστη, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο διακλαδικός ή διατομεακός δεσμός έχει πολύ ευρύτερη λειτουργία και σημασία όπως ε, τη διαφάνεια της αγοράς, την έρευνα, τη διαμόρφωση όρων. Επομένω να μπορούν να συνεπάρχουν και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να συνεπάρχουν. Και αυτό που είπε ο Γερμανός εκπρόσωπος εκείνη την ε, ημερίδα ήταν ότι λόγω της δομής των συνεταιρισμών στην ε, Γερμανία δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι θα χρειάζονταν οι διατομεακοί οργανισμοί. Γιατί θεωρήθηκε ε, αρχικά ότι θα τους κάλυπταν οι συνεταιρισμοί. Και όμως όχι. Πάλι από τη Γερμανία βλέπουμε ότι δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα τα δύο. Απλώς πρέπει να προσδοριστούν τα όρια των ρόλων. Άλλο κάνει ο συνεταιρισμός και άλλο, πιστεύω εγώ, ο διατομιακός οργανισμός. Και κάτι άλλο. αν υπάρχει διάκριση μεταξύ βορρά και νότου, αν υπάρχει ένα χάσμα. Νομίζω ότι η Γαλλία δείχνει με το παράδειγμα της αλλά και άλλες χώρες, Ουγγαρία, Ρουμανία, ότι υπάρχει, ότι δεν είναι τέτοιο το χάσμα. Η ε, Ουγγαρία, η Δανία, παραδείγματι, δεν έχει δείξει τέτοιο ενδιαφέρον. Και εδώ έρχομαι στο άλλο ζήτημα που επισημαίνεται, που είναι η επαγρύπνηση, η ευαισθητοποίηση. Εμείς διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μεγάλη επιθυμία για συμμετοχή με αυτή την ημερίδα της 24ης Μαρτίου. Ε, είδαμε ενδιαφέρον, αλλά η ευαισθητοποίηση δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Ας το πούμε αυτό. Θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να σταθούν και να στηρίξουν αυτό το έργο γιατί μπορεί να γίνει πιο εύκολα ή πιο δύσκολα αυτή η διαδικασία. Μπορεί κανείς να εξηγήσει τα πράγματα απλά στον παραγωγό του, στη γλώσσα του ή να μην το πράξει. Και άρα υπάρχει σημαντική, σημαντικό περιθώριο δράση από πλευρά μα και θέλουμε να ακούσουμε τι δικέ σα απόψει, αλλά μην τα φορτώνουμε και όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καλλιεργήσει και να προωθήσει εκείνη μόνο αυτό το σχέδιο. Και κάτι άλλο Οι διατομεακέ οργανώσει βεβαίω μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλυσίδα τόσο το καλύτερο όντως. Και όταν μιλούμε με διατομεακέ οργανώσει, πολλέ που είναι σύντομε, ε, μας λένε τι κρίμα που δεν έχουμε μεγαλύτερη έκταση περισσότερου εκπροσώπου τομέων. δεν εμπόριο παραδείγματι. Που σε ένα βαθμό εντάχθηκε. Άρα κάτι μπορεί να γίνει. Από την άλλη, αυτό που μπορώ να δώσω εγώ σαν απάντηση είναι ότι εάν ο διατομιακός οργανισμός θεωρηθεί ότι δεν αφορά μόνο τον ε, γεωργό, αλλά ολόκληρο τον τομέα, τότε μπορούμε να έχουμε μεγάλο κέρδος σε προσθέμενη αξία. Ευρωπαϊκός διατομιακός οργανισμός που ρώτησε κάποιος. Υπάρχει κανονισμός το 2016 που προβλέπει τη δυνατότητα αυτή. Μιλούμε για δια, ε, διεθνικούς διατομεακούς οργανισμούς, όπως αυτός ε, που φορά τα καπνά στην Ιταλία. Η σχετική νομοθεσία δηλαδή προβλέπει τη δυνατότητα. Από την άλλη, αν μιλούμε για επέκταση κανόνων ή τελών, πώς θα γίνει αυτό σε ένα εθνικό σύστημα καταπιστεύματος. Γιατί ναι, μπορεί να το κάνετε στη Γαλλία. Αλλά αν θέλετε να πάτε στην Ιταλία και να δείτε ε, για το πεπόνι το δικό σας τι τέλη καταβάλλονται στην Ιταλία θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Άρα ναι, μπορεί να υπάρχουν διεθνικοί οργανισμοί. Ε, και για να ολοκληρώνω, ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός ήταν ακριβώς τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά όργανα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι κανόνε περί του ανταγωνισμού, όπως είπαν κάποιοι, ο κύριος Νίκολσον, βεβαίως θα πρέπει να είναι σαφής, σε αυτό συμφωνούμε, το δείχνει μελέτη, ότι όσο πιο σαφής είναι η στόχοι και τα καθήκοντα του καθενός, τόσο καλύτερα. Από την άλλη δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης με το άρθρο 210 του κανονισμού για την ενιαία αγορά έχει ορίσει τους ε, κανόνες. Λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν προστασίες, εκμεταλλεύσεις προστασίες θέσει κτλ. Άρα ήταν ξεκάθαρο για τον Ευρωπαίο νομοθέτη ότι πλαισιωμένο αυτός ο διατομιακό οργανισμός μπορούσε να φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά ότι έπρεπε να προσδοριστεί το πλαίσιο. Ελπίζω να απάντησα. Σα ευχαριστούμε. Καταρχήν ε, να ευχαριστήσω θερμά και να εκφράσω τη χαρά μου και το θαυμασμό μου για την ε, έκθεση αυτή. Είναι ε, σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι εξίσου το εργαλείο αυτό σε όλες τις χώρες. Ε, και φυσικά εξαρτάται και από τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου, του κάθε τομέα. Και ακριβώς πρόκειται για διακλατή οι διατομιακέ οργανώσεις, ίσως μερικές φορές σε μερικά σημεία είναι ανταγωνιστικές προς τους συνεταιρισμού. Και ίσως γι' αυτό δεν ε, έγινε αποδεκτή η παρουσία της, δεν αναπτύχθηκαν δεόντως σε μερικές χώρες. Επίσης θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν αυτή θα είναι η απάντηση σε κάποιες κρίσεις, ιδιαίτερα με την ε, ε, κατάργηση των ποσοστώσεων όπω συνέβη στη ζάχαρη, στο γάλα ή στον τομέα των καπνών. Ε, μιλήστε και για το υλικό, τα έγγραφα αυτής της διάσκεψης. Μπορούμε να τα λάβουμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμα για μας τα έγγραφα αυτής της ε, διάσκεψης. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το περιλάβουμε αυτό και στη συζήτηση με τους εθνικούς βουλευτές. Γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την αλυσίδα τροφίμων. Ε, θα ρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και περιμένουμε την επόμενη ανάλυση και παρουσίαση Αυτά. Αύριο ξεκινούμε στις 9 με τις ψηφοφορίες. Μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ε, ψηφοφορίας. Έχουμε πολύ πιεσμένο και φορτωμένο πρόγραμμα γιατί ε, δεν θα έχουμε το απόγευμα συνεδρίαση. Οπότε να είστε όλοι παρόντες από τις 9 να ξεκινήσουμε αμέσως με τις ψηφοφορίες. Καλό σας απόγευμα και ραντεβού αύριο το πρωί.